Uh, dear colleagues, I would like to open the, uh, the meeting um, and I would like to inform you that... Uh, Καλημέρα, λέει Πρόεδρος. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι μεταδίδεται από το Ιντερνετ η συνεδρίασή μας και όσον αφορά το πρώτο θέμα έχουμε την έγκριση της σημερινής διατάξεως η οποία σας έχει διαβαστεί στις 22 Ιανουαρίου. Αν δεν έχετε ενστάσεις θεωρώ ότι η μέρη διάταξη εγκρίνεται και τώρα για να κάνουμε τις ανακοινώσεις της Προέδρου και θέλω να ζητήσω ε, η Βέρμπα να μας πει για αυτό το διορθωτικό έγγραφο. Οπότε πάμε στο 3 κατευθείαν, δηλαδή την έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Και σας ενημερώνω ότι έχουμε ε, τα πρακτικά Δευτέρα Ιουλίου, 1 Οκτωβρίου, 10 της Οκτωβρίου, όλα αυτά ε, είναι διαθέσιμα και σύμφωνα με την πάγια πρακτική θεωρούμε ότι εγκρίνονται εάν δεν έχουμε ενστάσεις μέχρι το τέλος αυτής της συνεδρίασης. Και τώρα πάμε παρακάτω στο 4 που είναι η ενημέρωση από πλευρά μου για το τι έγινε σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις του Brexit την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, αμέσως μετά την προηγούμενη δική μας συνάντηση και σας ενημερώνω ότι είχαμε αυτή την διευθύνουσα ομάδα BSG στις 23 Ιανουαρίου και τότε συζητήσαμε το πώς ε, έχουν τα πράγματα, ε, πώς έχει κατάσταση για το Brexit και αυτό λαμβάνω ε, με υπόψη της ψηφοφορίας σε σχέση με την Πρωθυπουργό κυρία Μέη στην Βουλή των ε, Κοινοτήτων. Ε, αυτά δημοσιοποιήθηκαν την 5η 24 πρώτο και σε αυτή την ε, δήλωση της Πρωθυπουργού ζητήθηκε από την, ε, από το, από την κυβέρνηση του ΕΒ να συνεργαστεί με όλους στην Βουλή των Κοινοτήτων, τόσο ώστε να απεμπλακεί το θέμα και ξανά ότι εμείς προσδοκούμε ότι θα υποβληθεί πρόταση από πλευρά Άγγλων για το πώς θα προχωρήσουμε. Επίσης, ε, είπαμε ότι η συμφωνία για την αποχώρηση δεν υπόκειται σε επαναδιαπραγμάτευση και επαναλάβαμε ότι πάγια υποστηρίζουμε ότι έχουμε ανοιχτό πνεύμα όσον αφορά τις μέλουσες σχέσεις μας με τον Εμμύριο Βασίλειο. Όμως ξεκαθαρίσαμε σε αυτή την ανακοίνωση ότι η κατάσταση όπως έχει τώρα κατατείνει περισσότερο στο να υπάρχει μια άτακτη αποχώρηση που δεν συμφέρει κανένα. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστεί από οποιασδήποτε ε, συγκεκριμένες ρυθμίσεις μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, στις 23 Ιανουαρίου έγινε μια συνάντηση, στις οποίες προείδευσε εδώ στο Κοινοβούλιο και αφορούσε το κατασκευαστικό φόρουμ. Οπότε και προσωπήθηκαν ε, διάφοροι κλάδοι της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας σε σχέση επίσης και με το Brexit. Και μας είπε για το πώς έχουν τώρα οι διεργασίες προετοιμασίας, ε, τι γίνεται από πλευρά επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για το Brexit, πώς θα γίνει επομένως ε, ο συντονισμός των εθνικών δράσεων προετοιμασίας και έγιναν ε, μακρές συζητήσει σε αυτό το φόρουμ και προέκυψε σαφω ότι όλοι είναι κατά του να έχουμε άτακτη αποχώρηση χωρί συμφωνία δηλαδή. Και ξεκαθαρίστηκε, ότι θα πρέπει να ξεβρεθεί μια λύση και ότι η βιομηχανία θα πρέπει να προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα και για αυτήν την ε, ε εκδοχή. Όπως όλοι γνωρίζετε, τι είπατε, λέει ο Πρόεδρος, συζητεί με τον Γραμματέα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω επίσης πως ελπίζουμε ότι η πρόταση της ε, κυρίας Μέπη επιδέχεται τροποποιήσεις και θα γίνουν τροποποιήσεις και ελπίζουμε ότι έτσι θα καταλήξουμε σε κάποια δημιουργική, επικοδομητική λύση. Αλλιώς, όπως το νησιό Μπαρνία, πάμε κατευθείαν για το σενάριο no deal, άτακτη δηλαδή αποχώρηση. Επίσης, να σου ό,τι γίνεται σχετικά με τη ε, διαδικασία της συνένεσης και σας υπενθυμίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Και έχουμε επίση αυτή την αναπομπή αυτή τη απόφαση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ε, αποχώρηση από πλευρά του Συμβουλίου προ το Κοινοβούλιο. Έγινε η αναπομπή αυτή τη διαδικασία ε, και βρείτε και κάποια επιστόλια που θα συνοδεύσει αυτή τη διαδικασία και είπαμε ότι το αίτημα της συνένεσης διαβάστηκε στο Κοινοβούλιο πριν την υπογραφή. Και θα ενημερωθούμε ευθύς αμέσω. Όταν δηλαδή πέσει η υπογραφή. Επίσης, στην τελευταία συνάντηση τη διάσκεψης των Πρόεδρων, δηλαδή, το ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος Ταγιάννη ότι θα ανακοινωθεί επισήμως αυτή η αναπομπή στην ε, ΑΦΚΟ κατά αυτήν την ε, σύνοδο αυτής της εβδομάδας. Και θα γίνει η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας την Πέμπτη, αυτή τη εβδομάδα Μετά την Ολομέλεια. Επίσης, θα υπάρξει ενημέρωση προ εσά όσον αφορά το πώ πάντα τα σε αυτήν την Η Μαρτίνα όμως έχει στήσει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν τη δήλωση της ε, ομάδα για τον Brexit τη περασμένη εβδομάδα ε, σύμφωνα με την οποία ε, εάν δεν υπάρχει backstop δεν θα υπάρξει συμφωνία αποχώρηση. Θα επικρατήσει λοιπόν το χάος στη Βουλή των Κοινοτήτων, που θα έπρεπε να ονομάζεται Βουλή του Χάου κανονικά. Θα συζητηθούν και οι τροπολογίες. Και είμαι σίγουρη πως όλοι γνωρίζετε πως αυτά γίνονται στο πλαίσιο κατηγοριών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαν να έρχονται δύο ταλίκες η μία πάνω στην άλλη και η μία από τις δύο θα πρέπει να κάνει πίσω. Διαφορετικά δεν θα αποφευχθεί η σύγκρουση. Κατηγορείται λοιπόν το Συμβούλιο και η Κομισιόν ότι παίζουν αυτό το παιχνίδι και κατηγορούμαστε και εμείς στη Βόρεια Ιρλανδία. Και ο Μάρτιν Μαγκίνες μας κατηγόρησε επίσης ότι παίζουμε αυτό το παιχνίδι Επίσης, η Βρετανία θα πρέπει να εφαρμόσει περίπου 600 ε, διατάξεις του ΠΟΕ, καθώς και ένα πλήθος άλλων κανονισμών σε περίπτωση αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ζήτημα ετοιμότητας και πρέπει να αρχίσουν να γίνονται πράγματα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν αρχίζουν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για ε, να μην έρθουν αντιμέτωποι με μία άτακτη αποχώρηση. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο ε, είχαμε δύο σημαντικές ειδήσει στην Ιρλανδία. Ένα συνέδριο με συμμετέχοντες που ανησυχούν πάρα πολύ για την απώλεια δικαιωμάτων μετά την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης μια εκδήλωση στα σύνορα. Στήθηκαν σκληρά σύνορα και μετά τα διέλυσαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο κόσμος λοιπόν στην Ιρλανδία, ειδικά στη Βόρεια Ιρλανδία, πιστεύει πως ε, αυτό δεν είναι παιχνίδι. Θέλει να πιστεύει πως είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να ε, διατηρηθεί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Πρωτού δώσω το λόγο στην ε, Μπάρμπαρα Σπινέλη, θα σας ενημερώσω λοιπόν πολύ σύντομα πως ίσως έχετε λάβει μια διόρθωση για την ε, ψηφοφορία της παρεσμένης εβδομάδα σχετικά με την έκθεση Σπινέλη για τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Υπάρχει ένα τεχνικό λάθος, το οποίο αν ε, δεν κάνω λάθος είναι αμεληταία σημασία και δεν επηρεάζει το περιεχόμενο το οποίο ψηφίσατε. Όμως οι σκιώδεις συμφώνησαν να ψηφίσουν στις πολιτικές ομάδες θα χρειαστεί λοιπόν να ψηφίσουμε την διόρθωση αυτή ως πρώτο σημείο στις ψηφοφορίες. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ πολύ, Ντανούτα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν για το διορθωτικό αυτό σημείωμα. ήταν σημαντικό για τη διαφάνεια. Και απαραίτητο, ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ενημερώθηκαν οι συντονιστές. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ λοιπόν Φτάνουμε στο τέλος των ανακοινώσεων και της ενημέρωσης για τον Brexit και θα περάσουμε στο σημείο 5 της υπηρεσίας διάταξης. Έχουμε τον κυβερνητικό τεταλμένο Γιώργια Τσιάμπα, Ευρωπαϊκό, ε, κυβερνητικό τεταλμένο λοιπόν της Ορμανικής Προεδρίας για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω κύριε Τσάμπα για να μας ενημερώσετε για τις προτεραιότητες της Ορμανικής Προεδρίας και για το πώς σκοπεύετε να συνεργαστείτε με την Επιτροπή ΑΦΚΟ τους ε, ερχόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χούπνερ. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ ως Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ρουμανίας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας. Είναι η πρώτη Προεδρία της ε, Ρουμανίας και θα αναφερθώ καταρχάς στις προτεραιότητές μας και το σκεπτικό πίσω από την ιεράρχησή τους και έπειτα θα ε, παρουσιάσω ορισμένα θέματα συνταγματικής φύσης με τα, για τα οποία συνεργαζόμαστε στενά με εσά. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αναλάβαμε την Προεδρία με μεγάλες φιλοδοξίες αλλά και ρεαλισμό και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Συνεργαζόμαστε λοιπόν επικοδομητικά έτσι ώστε να προχωρήσουν οι φάκελοι όσο το δυνατόν περισσότερο, διατηρώντας όμως την ενότητα και ενισχύοντας τη συνοχή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αποφασισμένοι λοιπόν να διασφαλίσουμε συνέχεια στο, στην ατζέντα της Προεδρίας και να το κρατήσουμε αυτό μέχρι το τέλος της εντολής μας. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν στηριζόμαστε στην δική σας στήριξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό εταίρος στην όλη διαδικασία και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί σε έναν επικοδομητικό διάλογο, ο οποίο θα οδηγήσει σε εξίσου επικοδομητική συνεργασία. Τους τελευταίους μήνες ο διάλογο μεταξύ της Ρουμανικής Προεδρία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ενεργός, ήταν επικοδομητικός και ελπίζω να διατηρήσουμε του τους ίδιους για τα θέματα με τα οποία θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικότερες προκλήσεις και για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Να πούμε ευθύ εξ αρχή ότι η πρώτη μας Προεδρία ξεκίνησε δυναμικά. Υπάρχουν πολύ δύσκολα θέματα, όπως το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το Brexit, οι ευρωεκλογές και η διαδικασία απολογισμού και προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, όλα αυτά ασκούν μεγάλη πίεση όχι μόνο στη δική μας Προεδρία αλλά και στις επόμενες. Και η Ρουμανική Προεδρία θα ε, προσπαθήσει να παίξει το ρόλο μεσάζοντα έτσι ώστε να επιληθούν τα θέματα αυτά, να εξασφαλιστεί συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν και επιλέξαμε την συνοχή ως κοινή ευρωπαϊκή αξία ε, για το σύνθημα της Προεδρίας μας. Χρειάζεται λοιπόν να προωθήσουμε και να στηρίξουμε τη συνοχή σε όλες τις, τις διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται ενίσχυση της συνοχής ε, της πολιτικής δράσης για να ενισχυθούν οι δεσμοί ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους πολίτες. Έπειτα χρειάζεται να ενισχυθεί η οικονομική διάσταση της συνοχής, διότι είναι η κινητήριος δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Τρίτον, ενίσχυση της ε, εσωτερικής διάστασης της συνοχής. Πρέπει να διατηρήσουμε την ε, σύγκληση και τις ε, θεμελιώδεις αξίες της ενιαίας αγοράς. Έχουμε λοιπόν καθορίσει τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Ε, τις έχουμε χωρίσει σε τέσσερις πυλώνες. Ασφαλέστερη Ευρώπη, Ευρώπη ως ισχυρός ε, παγκόσμιος παίκτης και Ευρώπη με ισχυρές αξίες. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε ε, τα σημαντικά έγγραφα, την δήλωση της Μπρατισλάβα, την, τη συμφωνία μάλλον της Μπρατισλάβα και τη δήλωση της Ρώμης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνοχή στο πλαίσιο του 18μηνου προγράμματος του Συμβουλίου, αλλά και της ε, τριπλής ε, προεδρίας με τη Φιλανδία και την Κροατία. Η προεδρία μας δεν έρχεται μόνο σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και η πρώτη από τις τρεις. Είμαστε λοιπόν ε, εμείς η χώρα η οποία θα πρέπει να καθορίσει τις προτεραιότητες για τους ερχόμενους 18 μήνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους τέσσερις πυλώνες, η Ευρώπη της σύγκλησης, η Προεδρία μας θέλει να διασφαλίσει σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να ε, υπάρχουν ίσες ευκαιρίες ε, για όλα τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε λοιπόν να στηρίξουμε την αύξηση του ανταγωνισμού, να αποδεχτούμε τις διαφορές και να προωθήσουμε την συνδεσιμότητα και την ψηφιοποίηση, να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα και ε, να παγιοποιήσουμε την βιομηχανική πολιτική. Δεύτερος πυλώνας, η Προεδρία μας είναι υπέρ μια ασφαλέστερη Ευρώπης, υπέρ τη αύξηση της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις ασφάλειας που απειλούν την Ευρώπη και τους πολίτες της. Τρίτος πυλώνας, η Ευρώπη ως ισχυρός ε, παγκόσμιος παίκτη. Στην ε, διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε κοινέ ε, πολιτικές, κοινή πολιτική γειτονίας και μια παγκόσμια στρατηγική η οποία θα διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τηρήσει τις διεθνείς της δεσμεύσεις. Τέταρτος πυλώνας, Ευρώπη με κοινέ αξίες. Είμαστε υπέρ της τόνωσης της αλληλεγγύης και της προώθησης πολιτικών για καταπολέμηση των διακρίσεων, για διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης σε άνδρες και γυναίκες. Επίση, την τόνωση τη συμμετοχή των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Η συζήτηση για την Ευρώπη θα είναι μία από τι ε, κυριότερε προτεραιότητε τη Προεδρία μα. Ελπίζουμε λοιπόν να είμαστε επικοδομητικοί και να προωθήσουμε μία συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ελπίζουμε στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ΑΦΚΟ ειδικότερα για τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Η Ρουμανική Προεδρία επίσης μέσω του Πρωθυπουργού της παρουσίασε τις ε, προτεραιότητές της και τόνισε την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης θα καθοριστούν οι προ... νέες προτεραιότητες περίπου τον Ιούνιο και εμείς ε, έχουμε κληθεί να ανταποκριθούμε στις... Ε, στην πρόκληση της ε, δημιουργίας λοιπόν των προτεραιοτήτων για το μέλλον της Ευρώπης. Στις 8 Ιανουαρίου, στη συνάντηση των Υπουργών Ιστορικών Υποθέσεων, συζητήθηκαν ήδη αυτά τα θέματα. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τον ε, διάλογο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για θέματα όπως το ψηφιακό θεματολόγιο και ε, άλλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογέ, η Σύνοδος του Συμπίου θα είναι ορόσημο για την Προεδρία μας και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία για να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας προς ε, την μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Η ατζέντα για τη στρατηγική αναμένουμε να εγκριθεί τον Ιούνιο κατόπιν συνένεσης και ελπίζουμε να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους επόμενους μήνες της Προεδρίας μας για να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε μέτρα που θα το πράξουν. Σε ό,τι αφορά τώρα την η ημερήσια διαταξή μα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα παραμείνει ψηλά στις προτεραιότητές μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα και όλα με, μετά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου τον περασμένο Δεκέμβριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τι ε, πολιτικέ δηλώσει 25η Νοεμβρίου, στόχο μα είναι να ολοκληρωθούν εγκαίρω οι διαπραγματεύσει για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δυστυχώ, όπω ε, γνωρίζετε, υπάρχουν αρκετά προβλήματα και αβεβαιότητα. Το Brexit, λοιπόν, θα πρέπει να ανέβει ακόμα ψηλότερες προτεραιότητές μας και για, και για να επιληθούν τα προβλήματα θα πρέπει να συνεργαστούν όλα τα θεσμικά όργανα. Είμαστε πεπισμένοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εργαστεί εξίσου αδιάκοπα για την εφαρμογή της συμφωνίας και ελπίζουμε να έχουμε τη στήριξή σας έτσι ώστε πριν το τέλος του Μαρτίου να εγκριθεί η συμφωνία. Τώρα, ας περάσω σε ορισμένα από τα θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή σας. Θα συνεχίσουμε την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει για τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες, ιδιαίτερα εν ώψη ευρωεκλογών. Δηλαδή, η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου και το ιδέσμι μέτρων για τις ευρωεκλογές. η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, το Μητρό Διαφάνειας, μεταξύ άλλων. Τώρα, οι μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δίκαιες και ελεύθερες ανεξάρτητες εκλογές είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Προεδρία μας. Επίσης, η νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ιδρυμάτων είναι εξίσου σημαντική και ελπίζουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις. Ελπίζουμε λοιπόν να εργαστούμε γρήγορα έτσι ώστε να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο η σχετική νομοθεσία και να τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Απρίλιο, πριν δηλαδή από τι ευρωεκλογέ. Σε ό,τι αφορά τώρα το μη νομοθετικό σκέλο τη δέσμη μέτρων για τι ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ, το Φεβρουάριο Έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες ε, συζητήσεις. Ήδη τον Ιανουάριο στην Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έχει συζητηθεί αυτό το θέμα καθώς και οι διάφορες πτυχές ε, διεξαγωγής των εκλογών. Είναι πολύ σημαντικό να συγχρονιστούν οι ε, ευρωεκλογέ ε, σε, όλες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνουν με πιο δίκαιο και ελεύθερο τρόπο. Να αποφύγουμε την χειραγώγηση όπως την τελευταία φορά και να δώσουμε στους πολίτες ε, την ε, δυνατότητα της ελεύθερης ε, της ψηφοφορίας κατά βούληση, χωρίς χειραγώγηση. Χρειάζεται λοιπόν ένα μέσο συνεκτικής επικοινωνίας και συντονισμός όλων των θεσμικών οργάνων για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δεν πρέπει λοιπόν μόνο να δίνουμε βάση στη στρατηγική αλλά και στους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να επικοινωνούμε με τους πολίτες ακόμα και για ίσονο σημασία θέματα, τα οποία όμως αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου ζήτησε να συνεχίσει η δουλειά για αυτό το θέμα ε, επόμενη συνεδρία είναι το Μάρτιο του 2019 και στις 5 Δεκεμβρίου είπα ότι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε τις προτεραιότητές της. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εγκριθούν εγκαίρως. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε προορατικοί, να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε να συμπεριληφθεί τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και η βιομηχανία και οι άλλοι κλάδοι στην προσπάθεια αυτή. Χρειάζεται λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα περιλαμβάνει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική διάσταση των ευρωεκλογών. Σεβόμενοι ταυτόχρονα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις 8 Ιανουαρίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συζητήθηκαν τα επίγοντα θέματα, γι' αυτό λοιπόν ε, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και τους ερχόμενους μήνες με τις προτεραιότητες ε, σχετικά με το σχέδιο δράσης. Όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ, είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης ε, της πληροφόρησης. Ενημέρωση των πολιτών και ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στις ε, παρεμβολές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Μητρό Διαφάνειας, ελπίζουμε οι διαπραγματεύσεις να συνεχίσουν με τρόπο επικοδομητικό. Είμαστε σίγουροι πως ε, θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Εμείς δεσμευόμαστε προς την έβρεση μιας ικανοποιητικής λύσης, ε, διότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη Ρουμανική Προεδρία. Θέλουμε λοιπόν να επαναλάβουμε την δέσμευσή μας για ε, επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Διότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Η μόνιμη αντιπροσωπεία μας στις Βρυξέλλες επίσης ε, ασχολείται ενεργά με το θέμα αυτό. Τώρα, έχει συζητηθεί και το non-paper, το οποίο αναφέρεται στην ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να βρουν κοινά σημεία και συνεχίζουμε την συνεργασία. Υπάρχουν όμως αρκετές ανησυχίες με τα κράτη-μέλη για ε, πολλά επιμέρους ζητήματα. Θέλουμε λοιπόν να συνεχιστεί ο διάλογος και να ε, οδηγηθούμε σε μια αποκριστάλλωση των θέσεών μας. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεχίσουμε το έργο της Αυστριακής Προεδρίας και να ε, έχουμε και εμείς αυτήν την επικοδομητική προσέγγιση, έτσι ώστε να συνεχίσουμε το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Τώρα, δεν μου φαίνεται πολύ ρεαλιστικό ε, το, ότι, το χρονοδιάγραμμα και δεν νομίζω να καταφέρουμε να επιτύχουμε μια λύση μέσα σε αυτό το τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον ε, διοργανικό διάλογο και θα ήθελα να ολοκληρώσω ε, τονίζοντας ακόμη μια φορά ότι η Ρουμανική Προεδρία, Προεδρία θα συνεισφέρει στην δρομολόγηση και ολοκλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ε, θεμάτων το πρώτο τρίμηνο της Προεδρίας της πριν τις ευρωεκλογές. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στα μη νομοθετικά ζητήματα, τα οποία όμως είναι εξίσου περίπλοκα και σημαντικά και η Προεδρία μας θα καταβάλει προσπάθειες για την δημιουργία συνένεσης στους τριμερείς διαλόγους και αναγνωρίζει φυσικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Η Ρουμανία λοιπόν δεσμεύεται να μεσολαβήσει στο Συμβούλιο έτσι ώστε να διευκολύνει τον ε, διάλογο. Ελπίζουμε λοιπόν ε, και στην δική σας επικοδομητική και προορατική προσέγγιση, όπως γνωρίζετε, χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση από όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά και τα κρατημέλη. Γνωρίζουμε πως είναι εξίσου σημαντικό για όλους να έχουμε θετικά αποτελέσματα ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουμε στις ευρωεκλογέ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, ιδιαίτερα στο ε, ιδιαίτερα δεδομένων των ευρωεκλογών. Αναμένουμε λοιπόν ε, θετικά αποτελέσματα, διότι αυτό το θετικό αποτέλεσμα είναι ουσιώδες έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρή φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία μετά τις ευρωεκλογέ, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε και Σάμπα για αυτή την πολύ αναλυτική παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας. Προφανέ ότι η Ρουμανία θα προσπαθήσει να βρει αποτελέσματα σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά και για μα, αλλά όπω πολύ σωστά είπατε έχουν σχέση και με την ποιότητα των ευρωεκλογών. Αυτό θα είναι μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο ω Ευρωκοινοβούλιο, αλλά ω Ευρώπη συνολικά. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους, ξεκινώντας από τους ε, εισηγητές των πολιτικών ομάδων, ξεκινώντας από το ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ κύριο Σεπφλίν. σα ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας. Είναι πάντοτε δύσκολο όταν ε, για πρώτη φορά μια χώρα αναλαμβάνει την εκπαιδευτική της Προεδρία του Συμβουλίου. Το γνωρίζουμε. Το πρώτο ζήτημα που αναφέρατε και που θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις ευρωεκλογέ είναι η κυβερνοασφάλεια. Θα ήθελα να μα δώσετε λίγε περισσότερε λεπτομέρειε πληροφορίε για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κυβερνοασφάλεια. Θα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και επίσης, θα ήθελα να μου πείτε, τι πιστεύετε εσείς, γιατί είναι ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση οι πολίτες, γιατί είναι τόσο εύπιστοι, γιατί με τόση ευκολία πιστεύουν ψέματα. Θα ήθελα να μου πείτε τις απόψεις σας για το θέμα. Αναφέρατε επίσης το ζήτημα της, των γειτονικών χωρών της ε, γειτονιά μας και θα ήθελα να μας πείτε, αν και δεν είναι άμεσα θέμα της ΑΦΚΟ, ε, τι πιστεύετε για την Σερβία. Πιστεύουμε, ο, πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας θα έχει πολύ σημασία, μεγάλη σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή και για πολλές άλλες γειτονικέ χώρες, όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία. Είπατε επίση ότι ότι θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι ακριβώς αυτό εννοούσατε. Δεν φαντάζομαι ότι θα ολοκληρωθεί ποτέ η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Αν ποτέ συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Για την ομάδα των σοσιαλιστών, Ραμόν Χαουρέκη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε και εκ μέρους της ομάδας των σοσιαλιστών, κύριε Υπουργέ. Έχω ορισμένε ερωτήσει για εσά κυρίω σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Μια και είπατε ότι θα είναι ένα από τα κεντρικά θέματα της ε, Ρουμανικής Προεδρίας. Πρώτα απ' όλα, εκ μέρου τη ε, ομάδα των Σοσιαλιστών. Θα πρέπει να, να σα διαβεβαιώσω ότι, έχουμε, ότι έχει η χώρα σα και οι ηγέτε τη ε, την πλήρη εμπιστοσύνη μα για να ηγηθείτε αυτή τη δύσκολη περίοδου έχουμε διαπιστώσει και τον επαγγελματισμό το, και επίσης την ε, αποφασιστικότητα που έχει δείξει η κυβέρνησή σας και την προσπάθεια που έχει καταβάλει για την ε, Προεδρία. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταλήξει σε μια σειρά εκθέσεων σημαντικές για την ενισχυμένη συνεργασία, για την διαφοροποιημένη ενοποίηση κτλ. Ε, είναι ζητήματα σημαντικά αυτά για τους πολίτες γιατί με αυτέ τι εκθέσει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων δίνει κάποιε γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ για το προ το που πρέπει να κινηθεί στο μέλλον η Ευρώπη. Και θα πρότεινα να αξιοποιήσετε τη σύνοδο του Σύμπιου για να εμβαθύνετε τη συζήτηση πάνω σε αυτέ τι ιδέε, και να ξεκινήσει και να, να, να τεθούν επιτάπητος αυτές οι βασικές ερωτήσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Χρειάζεται μια πολιτική συζήτηση, κύριε Υπουργέ, για, τις μεγάλες, για τα μεγάλα αυτά ζητήματα για το μέλλον της Ευρώπης τους επόμενους μήνες και, αργότερα. Ε, κατά την άποψή μου πρέπει να καταπολεμήσουμε τον λαϊκισμό, τους διάφορους, τον αντιευρωπαϊσμό, αντιευρωπαϊσμό και τους διάφορους άλλους ισμούς που μας κατατρέχουν. Και για να το καταφέρουμε αυτό, ε, ο καλύτερος τρόπος είναι να εκθέσουμε ξεκάθαρα στους πολίτες μας ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα, τα μεγάλα διλήμματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Και να αξιοποιήσουμε τις ευρωεκλογέ για να εκφράσουν οι πολίτες την άποψή τους για την Ευρωπαϊκή Ενωπήση. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρομαι και σε αυτές τις συγκεκριμένες εκθέσεις, οι οποίες θα εγκριθούν και από την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου, για αυτά τα σημαντικά ζητήματα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο. Θα ήθελα να με ενημερώσετε τι σκοπεύει να κάνει η ε, Ρουμανική ε, Προεδρία για το ζήτημα των ευρωεκλογών σε σχέση με το Brexit, δηλαδή τι θα συμβεί με τους ευρωβουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, τι λύσεις έχετε σκεφτεί για να σεβαστούμε από τη μια το δικαίωμα που θα έχουν οι Βρετανοί πολίτες να ψηφίσουν εάν ακόμα δεν έχει συμβεί το Brexit. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και θα περιμένουμε από την πλευρά της Ρουμανικής Προεδρίας να δώσει μια κατεύθυνση σε αυτή τη συζήτηση που θα χρειαστεί. Τρίτον, θα ήθελα συγκεκριμένα να μας πείτε εάν έχει αποφασίσει η Ρουμανική Προεδρία να εγκαταλείψει την συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί ε, έχω την εντύπωση, ε, δυστυχώς, ότι δεν υπάρχει πλέον ένα πολιτικό περιθώριο για να διαπραγματευτούμε τους προτεραιότητες και την κατανομή των πόρων στο MFF. Αλλά θα χρειαστεί να υπάρξει μια συμφωνία. Και Έρχομαι τώρα σε ένα ζήτημα που είναι πιο συγκεκριμένο ε, ε, αρμοδιότητα της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Είναι το δικαίωμα ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δημιουργεί διερευνητικέ επιτροπές. με, αυτό το, με αυτή την προσπάθεια, με αυτή τη συζήτηση μάλλον, προσπαθούμε να δείξουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ του Συμβουλίου ε, στη συζήτηση του θέματος αυτού, δυστυχώς. Αυτό το, το εκθέτουμε, το εκφράζουμε με την έκθεσή μας. Προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο η ΑΦΚΟ να αναδείξει το θέμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, να ξαναθέσει το θέμα στο Συμβούλιο. Μιας λοιπόν και θα είστε προεδρεύουσα χώρα στο Συμβούλιο, σας ζητώ να λάβετε υπόψη σας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερο ενοχλημένο από αυτήν την κατάσταση, γιατί θεωρούμε ότι έλειψε η ε, σωστή συνεργασία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα θεσμικά όργανα σε αυτό το θέμα, στο δικαίωμα διερεύνησης. Ευχαριστούμε κύριο Σπρέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε κύριε Υπουργέ. Ιδιαίτερα ευτυχή που σας βλέπω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σα εύχομαι καλή επιτυχία και εσάς και στους συνεργάτες σας. Δυο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με τη σύνοδο του Σύμπιου, στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Όταν αποφασίστηκε να διοργανωθεί αυτή η σύνοδος του Σύμπιου, υπήρχε μια σχετική αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχώρησή του. Και σε αυτό το πλαίσιο λέγαμε και σκεφτόμασταν ότι θα έχουμε μια δυνατότητα στη Σύνοδο του Σύμπιου να συζητήσουμε οι υπόλοιποι ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλάξαν όμως τα πράγματα και τώρα υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με την ε, Συμφωνία Αποχώρησης. Υπάρχει η πιθανότητα καθυστέρησης του Brexit. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ, μήπως, πρέπει, μήπως χρειάζεται και τι πιστεύετε εσείς να, να αλλάξουμε την ε, ημερήσια διάταξη της συζήτησης που θα γίνει στο ΣΥΠΙΟΥ. Αν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου γίνει χωρί συμφωνία, άτακτα, αυτό σίγουρα θα αλλάξει την συζήτηση στο ΣΥΠΙΟΥ. Δεν θέλω να μου πείτε την άποψή σας γι' αυτό. Δεύτερον, ε, το ανέφερε και ο κύριος πλήν ήταν μια συζήτηση στην οποία, oh, στην οποία μας εκπροσωπούσε και η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας. Μιλώ για την πρωτοβουλία των πολιτών. Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίθηκε και από την Ολομέλεια το Δεκέμβριο και θα αρχίσουν να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο. Και αυτό το νέο σύστημα για την πρωτοβουλία των πολιτών προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος θα έχει την δυνατότητα να επιλέγει το ελάχιστη, την ελάχιστη ηλικία ε, των πολιτών που μπορούν να συνυπογράψουν μια τέτοια πρωτοβουλία από Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή όταν θα είναι 16-18 χρόνια. Υπό αυτή την έννοια δηλαδή έχει αποσυνδεθεί η ελάχιστη ηλικία για να συμμετάσχει στις εκλογές από την ελάχιστη ηλικία για να συνυπογράψει μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Και θα ήθελα να μου πείτε κύριε Υπουργέ, εάν πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα αυτό. Είναι καλή ιδέα να μπορούν οι 16χρονοι να ε, εμπλέκονται στα πολιτικά έτσι. Τώρα προσωπικά εγώ θα πίστευα ότι οι 16χρονοι θα έπρεπε να είχαν και δικαίωμα ψήφου, αλλά ξέρετε όταν το πρότεινε αυτό στη Ρουμανία δεν έτυχε καλή υποδοχή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, είστε ανοιχτοί, είστε υπέρ αυτή τη συμμετοχή των ε, νέων παιδιών των 16χρονων στον πολιτικό διάλογο. Ευχαριστούμε. Γιατί Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Είναι η πρώτη φορά που η Ρουμανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είναι μια από τις σημαντικότερες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εδώ εξετάζεται το κατά πόσον η νομοθεσία που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο μέλλον. Ε, και σίγουρα τα τελευταία χρόνια ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεχτεί διάφορα πλήγματα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, από τα προβλήματα με τη μετανάστευση, από το Brexit και έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα για το ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης. Έχει ακουστεί επίσης και η ιδέα της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων. Κατά την άποψή μου, είναι σοφή η επιλογή που έκανε η Ρωμανική Προεδρία να τονίσει το ζήτημα της συνοχής, της ενότητας στην Ευρώπη, γιατί κατά την άποψή μου ότι είναι αυτός ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουμε το μέλλον που επιθυμούμε στην Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το πρόβλημα του Brexit. Είναι αλήθεια ότι δεν, δεν, δεν στάθηκε δυνατό να επικυρωθεί η Συμφωνία Αποχωρήσης από τη Βουλή των Κοινοτήτων και αυτό δημιουργεί μια σειρά προβλήματα ανάμεσα σε αυτά και ένα πρόβλημα με τις ευρωεκλογέ. Ένα άλλο ζήτημα που εγώ θα ήθελα να θέσω είναι το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να έχουν ελευθερία μετακίνησης και το δικαίωμά τους να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Εφόσον λοιπόν δεν έχει ακόμα εγκριθεί η συμφωνία αποχώρησης, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ε, προστατέψουμε αυτά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Τέλος. Κάθε φορά που συζητούμε για το μέλλον της Ευρώπης, συζητούμε και για τον εξτρεμισμό, για τον λαϊκισμό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θεωρήσει, έχει αναγνωρίσει την κίνδυνο που υπάρχει εδώ. Θα ήθελα να μου πείτε τι προβλέπει να κάνει για αυτά τα ζητήματα η Ρουμανική Προεδρία. Αυτό, αυτός, αυτοί οι διαφορετικών ειδών εξτρεμισμοί θέτουν σε κίνδυνο ε, και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά και το μέλλον των ε, χωρών μας. Νομίζω αρκετέ ερωτήσει σα έθεσα. Σα εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στην Προεδρία σα. Μερσέντε, θέλετε το λόγο. Θέλει κάποιο άλλο συνάδελφο το λόγο. Να προσθέσω κι εγώ κάτι, λέει η κυρία Χούμπλερ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε. Ιδιαίτερα τη συνεργασία που είχαμε για την αλλαγή των κανόνων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, τις αλλαγές που επιτύχαμε σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, ε, αλλαγές στην νομοθεσία που τις, εμείς τα μέλη του Κοινοβουλίου θεωρούσαμε πολύ σημαντικά. Ε, αναφερθήκατε ε, στην σημασία που έχει η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Εμείς προβλέπουμε τον Απρίλιο να οργανώσουμε μια διακοινοβουλευτική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Είπατε ότι θα εγκρίνει Προβλέπετε τον Ιούνιο μια στρατηγική για το θέμα του Συμβούλιο. Επί τη βάση της Οργανικής Συμφωνίας πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια από κοινού συνεργασίας και μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, όχι μόνο κατά τη διάρκεια ενός έτους, αλλά σε πολιετές επίπεδο και για πρώτη φορά καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια κοινή δήλωση για τη στρατηγική, την πολιετή για το μέλλον της Ευρώπης. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, αυτό το ζήτημα δεν θα το ε, εξετάσει η Προεδρία σας, αλλά η επόμενη. Πάντως, θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε έτοιμοι για να καταλήξουμε σε κοινή δήλωση, δηλαδή. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε στο Συμβούλιο ότι θα είναι κοινή η δήλωση, στην οποία δηλαδή θα τη συνυπογράφει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή τη δήλωση για το μέλλον της Ευρώπης. Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς πώς βλέπετε την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη συζήτηση, για παράδειγμα στη Σύνοδο στο ΣΥΠΙΟΥ, δεδομένου μάλιστα ότι θα βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Παρά την προεκλογική περίοδο όμως πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο να έχουμε μια ε, συμμετοχή στην ε, Σύνοδο του ΣΥΠΙΟ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Σας δίνω τώρα το λόγο για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Υπουργός. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση που έθεσε ο κύριος Σόπφλεν για την κυβερνό ασφάλεια Είναι θέμα ε, των αποφάσεων του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Εμείς έχουμε καλέσει τα εξεκράτη που ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία στα περιθώρια του Συμβουλίου εκείνου για τις ε, τιμίες εκλογές, ούτως ώστε να υπάρξει νομοθεσία για κυβερνοασφάλεια. Ε, πρόκειται για Πρόκειται για αυτούς τους κανόνες, rules of attribution, για το τι κυρώσεις επίσης θα επιβάλλονται σε περίπτωση που κάποιος ε, παρένδε εκλογέ στην ε, Ευρώπη. Τα είπαμε αυτά στα συμπεράσματα του Φεβρουαρίου. Τώρα όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συζητήσαμε και την παραπληροφόρηση και το πώς η Ευρώπη θα επικοινωνεί καλύτερα. Όταν αφήνουμε κάποιο κενό, το κενό αυτό θα πληρωθεί κατά κάποιο, θα συμπληρωθεί από αυτές τις ψευδείς ειδήσει. Ε, Επομένω χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία ε, στην Ευρώπη και για την Ευρώπη και έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε τι γίνεται ε, με όλες αυτές τις ψευδείς ειδήσει, όλα αυτά τα ψέματα που λέγονται για την Ευρώπη και για τα θεσμικά όργανα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε το θέμα να το αντιμετωπίσουμε ε, στα πλαίσια μιας σφαιρικής προσέγγισης της καλύτερης επικοινωνίας ε, και ε, βέβαια για την πολιτική γυρνίαση έχουμε φυσικά το θέμα ως προτεραιότητα γιατί και εμείς περάσαμε από την διαδικασία της διεύρυνσης που μας βοήθησε στην ανάπτυξη η νέα αγορά που μας έκανε ισχυρότερους. Και εμείς αποκτήσαμε την εμπειρία της προσχώρησης, οπότε ε, βεβαίω και προτιθέμεθα όλα αυτά να τα μοιραστούμε με τις χώρες που προσεγγίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε και αυτή την εκδήλωση της Προεδρίας για τα Δυτικά Βαλκάνια, είχαμε την συνάντηση κορυφής των νέων και επιστώσαμε η... το ρόλο της νεότερης ε, γενιάς συμφωνίες, συζητήσαμε για την συμφιλίωση, συζητήσαμε για προσέγγιση Γαλλίας-Γερμανίας, είπαμε πόσο σημαντική είναι η παρέμβαση των νέων σε αυτό και για τα Δυτικά Βαλκάνια όσον αφορά την συμφιλίωση και όσον αφορά το ότι θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας την προϊστορία που υπάρχει. Ε, επίσης, Θα πρέπει να υπάρχει η επόμενη στρατηγική θεματολογία που δεν πρόκειται να ολοκληρώσει την συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά πρόκειται να διαμορφώσει τις καθεντήρες γραμμές για την επόμενη πενταετία. Επομένως, είναι σημαντικό να αποκρισταλώσουμε κάποιες αρχές, αυτές επί των οποίων όλοι συμφωνούμε και ο καθένας να έχει όσο Ευρώπη θέλει και να μην έχουμε διαφορές, μην έχουμε όμως και Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Και όλα αυτά στο επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο να παγιωθούν και έτσι να διαμορφώσουμε την ε, προβληματική για το μέλλον για μια Ευρώπη που θα έχει τις ελάχιστες κατευθυντήριες σύμφωνα με το στρατηγικό θεματολόγιο τώρα όσον αφορά ε, το χρονοδοτικό πλαίσιο είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας αυτό το ε, χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να πετύχουμε τα σκοπούμενα αποτελέσματα. Ε, γιατί αν δεν πετύχει, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα φύγουμε. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό ε, αυτό να συζητείται σε κάθε Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο Θα πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο των προηγουμένων ε, προεδριών, των καλών πρακτικών για το πώς θα λειτουργεί το Συμβούλιο και να χωνέψουμε ό,τι έχει επιτευχθεί. Τώρα, όσον αφορά το, τα θέματα στρατηγικής, τακτικής, θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε όσον αφορά τον Box και όσον αφορά τις νομοθετικές πράξεις ανά τομέα, ανά κλάδο. Χρειάζεται βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια με τη νέα καταληκτική ημερομηνία δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια σα ίσα, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αλλιώς ποτέ δεν θα τηρηθεί καμία προθεσμία όσον αφορά τουλάχιστον την τρέχουσα θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας και τα συζητούμε διμερώς με τα κράτη-μέλη. Τα συζητούμε και στο Συμβούλιο. Οπότε γι' αυτό σας λέω, αναμένεται να σημειωθεί πρόοδος. Και αυτό σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να το προχωρήσουμε πιο γρήγορα γιατί θα χάσουμε κάποιες προθεσμίες πριν τον επόμενο προϋπολογισμό. Τώρα, όσον αφορά το δικαίωμα έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι και η Αυστριακή Προεδρία, μου επιτρέπετε να το πω, αλλά και οι πιο παλιέ ε, συμμετέσχουν σε αυτού του είδους την ε, ε, ευρία ανταλλαγή απόψεων και με επικοδομητικό τρόπο. Και εμείς θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Είχαμε ήδη κάποιες αντίσεις της ομάδας εργασίας και σας ότι έτσι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα για αυτό το περίπλοκο θέμα. Συμφωνούμε με το στόχο σας ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος. Τώρα, γι' αυτό πρώτος ο κύριος Πρέντα για το Συμπίου. Και για το Brexit. πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για τον Brexit. Ακόμα περιμένουμε να διευκρινίσει τις θέσεις της, τις προθέσεις της με συγκεκριμένες προτάσεις η Βρετανική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να κινηθούμε πιο γρήγορα για τα κατεπήγοντα μέτρα. Προς τα εκεί κινήθηκε το Συμβούλιο. Και κατόπιν θα τα συζητήσουμε και με εσάς. Οπότε σε επίπεδο κρατών μελών ε, γίνονται προσπάθειες και θα πρέπει τα κρατημέλη να νομοθετήσουν σχετικά. Βεβαίω και θα πρέπει να επιδείξει και καλή πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και στα θέματα της επιτροπολογίας, ε, γιατί και εκεί κάποια θέματα θα πρέπει να ρυθμιστούν σε αυτό το επίπεδο. Επίση έχω δεχθεί διαβεβαιώσεις προσωπικά από τον Βρετανό Υπουργό όσον αφορά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν θα φυγούν στο σενάριο της άτακτης αποχώρησης. Ήδη η Βρετανική κυβέρνηση έχει λάβει κάποια σχετικά μέτρα. Ήδη είχαν ξεκινήσει πιο πριν και τώρα υπάρχει εφαρμογή όσων, και υλοποίηση όσων είχαν ε, υποσχεθεί. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί έγκαιρα η συμφωνία για την αποχώρηση. Ε, και φυσικά τα κατεπίγοντα μέτρα αφορούν την περίπτωση που δεν θα υπάρχει συμφωνία. Βέβαια, όσο περισσότερη βιότητα υπάρχει, όσο περισσότερη βιότητα και όσο περισσότερα τα πράγματα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, τόσο πιο σημαντικά είναι αυτά τα μέτρα. Άρα, συνεχίζουμε να υπολογίζουμε στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει η επαύριον. Τι θα προκύψει από πλευράς Λονδίνου. Τι θα μας πει η Βρετανική κυβέρνηση. Καλόπιστα. Θα τα ακούσουμε. Πώ υπάρχει η πολιτική δήλωση, επί τη οποία έχουμε συμφωνήσει. Τα συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο και σύμφωνα θα, σύντομα θα έρθει και η σειρά ειδική να συμφωνήσετε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τώρα. Άλλο. Για την πρωτοβουλία των πολιτών και για την νεολαία. Όσον αφορά την πρωτοβουλία, προσπαθήσαμε στην Προεδρία να την διεκπαιρεώσουμε, να την προωθήσουμε και για, ακριβώς για τους νέους και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια από τους νέους πρέσβες σε συνεργασία με τη UNICEF και έτσι ε, να εμπλακεί στα ευρωπαϊκά πράγματα, σε ευρωπαϊκές υποθέσεις η νεολαία και βέβαια είναι και το θέμα του να ληφθεί απόφαση για το ηλικιακό όριο. Αυτό όμως είναι εθνική αρμοδιότητα. Δεν έχουμε επ' αυτού κοινοτική αρμοδιότητα κάποιου συγκεκριμένο για το θέμα του δικαιώματος του εκλέγην των νέων. Ό,τι φέρει καλύτερη επικοινωνία στην Ευρώπη, εμείς το ενθαρρύνουμε. Να ενθαρρύνουμε. Δηλαδή τις νεότερες γενιές. Να τις θωρακίσουμε από την παραπληροφόρηση σχετικά με την Ευρώπη. Να τους ενημερώσουμε για τα πλέον εκτήματα της Ευρώπης. Είναι θωρακισμένοι βέβαια έναντι αυτών των θεωριών ότι η Ευρώπη είναι κακή, ότι δεν έχει καμία προσθέμενή αξία για τους νέους. Η Ευρώπη βοηθάει για την έξοδο, την κρίση, για ανάπτυξη, για απασχόληση. Η ανεργία των ε, νέων ήταν ε, κορυφαίο θέμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ταχύτατα. Γιατί αλλιώς θα έφερνε απογοήτευση που δύσκολα αντιμετωπίζεται. Άλλο. Κυρία Ταπαρντέλ. Ναι, ναι, η σύνοχη είναι πολύ σημαντική. Είναι η έκφραση και η υλοποίηση της ενότητας. Και επίσης είναι η έκφραση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της ε, ενίας αγοράς. Ε, γι' αυτό δεν μπορεί να έχουμε επιλεκτική προσέγγιση. κινητικότητα, ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε διαφοροποιημένη προσέγγιση σε σχέση με τις άλλες τρεις θεμελιώδες ελευθερίες της αγοράς. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Ε, γι' αυτό και είναι σημαντική συνοχή. Αλλά αν θέλουμε να δείξουμε την ενότητα και την αποφυγή της διακρίσεων, ναι, αυτό θα βοηθήσει το ευρωπαϊκό όραμα θα βοηθηθεί και η καταπολέμηση του λαϊκισμού. Άρα να μιλούμε για το τι εκπροσωπεί η Ευρώπη, για τα επιχειρηματά της. Άρα εδώ έχει σχέση η πρωτοβουλία της Προεδρίας μας για καλύτερη επικοινωνία. Δεν θα πρέπει να ασχολούμεθα με ζητήματα που δεν απασχολούν τον κόσμο. Ούτε θα πρέπει να ασχολούμαστε με πάρα πολλά. Θα πρέπει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δούμε τι έχει καταφέρει ούτω ώστε η ζωή του Ευρωπαίου να είναι ευκολότερη. Διαπιστώνετε τι έχουμε καταφέρει. Όταν ε, ρίχνουμε μια ματιά για τις συνέπειες ε, της ε, έφτακτης ή άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Άρα θα πρέπει κανείς να σκεφτείτε καλά τι λέει για την Ευρώπη όταν αποφαίνεται για το πόσο αξίζει η Ευρώπη, πόσο ενώνει τον κόσμο, πόσο κάνει τον κόσμο να έχει μια αίσθηση του ανήκειν στην ίδια οικογένεια. Τώρα όσον αφορά τις ε, διοργανικές ρυθμίσεις, το διοργανικό πλαίσιο για καλύτερη νομοθεσία. Ήδη αυτό και άρχισε μας απασχολεί. Και υπάρχει κάποια άνηση, ασύμετρη πρόοδος, γιατί σε κάποιους τομείς έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε σε άλλους τομείς λιγότερο. Όμως, θα πρέπει να χωνέψουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος. Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το στόχο. Έτσι, θα διαμορφώσουμε και το τι θα γίνει σε επόμενες προεδρίες, όχι μόνο στη δική μας, τι σχέσεις μας τις σχέσεις Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, στο μέλλον κλπ. Άρα θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδο και καταλαβαίνουμε πολύ καλά βέβαια ότι η σημειακή πρόοδος δεν σημαίνει ότι διεκπαιρεώθηκαν όλα, αλλά τουλάχιστον είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω κάλυψα τα πάντα. Η πρόοδο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά όλα τα θεσμικά όργανα συνεχίζουν τη δουλειά και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα γίνει συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και για άλλα λιγότερο σημαντικά θέματα. Σας ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας, την πρώτη Προεδρία της Ρουμανίας. Ξέρω πως έχετε άριστο επιτελείο, που ασχολείται με την Προεδρία, γι' αυτό λοιπόν καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Σας ευχαριστώ όλους που με ακούσατε. Yeah, Yes, we are Thank you very much. Thank you very much. Great work. Um, dear colleagues, we continue the meeting. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ραμόν, συνεχίζουμε. Ίσως θυμάστε ορισμένοι ότι είχαμε ζητήσει από το Τμήμα Πολιτικής για τα δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις να ε, συντάξει μία μελέτη σχετικά με το ενωσιακό πλαίσιο για την επιβολή του σεβασμού στο κράτος δικαίου και στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ένωσης. είχαμε κατευθυνθεί από τις εξελίξεις για αυτά τα θέματα τα τελευταία χρόνια, όμως ε, νομίζω πως έχουμε κάνει αρκετά βήματα σχετικά με ε, τον εντοπισμό των τροτών σημείων στις συνθήκες και στο νομικό μας πλαίσιο. Η μελέτη λοιπόν αυτή νομίζω και ελπίζω ότι θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει στο έργο μας. Έχουμε λοιπόν μία παρουσίαση σήμερα, ε, η οποία θα μας ενημερώσει και για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη, ε, από καθηγητές συνταγματικού δικαίου, τον ε, καθηγητή Diego Λόπες Γκαρίδο από το Πανεπιστήμιο της Καστίγια Λαμάντσα και τον καθηγητή Αντώνιο Λόπες Καστίγιο από το Αυτόν Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Θα δώσω λοιπόν το λόγο και στους δύο καθηγητές. Η γραμματεία δεν με ενημέρωσε για πόση ώρα μπορείτε να μιλήσετε, μάλλον για 10 λεπτά έκαστος, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Κατόπιν θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Κύριε Καρίδο, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ τους βουλευτές της Επιτροπής σας. Ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε, τον Λόπεθ Καστήλιο και τον υποφαινόμενο και μας αναθέσατε αυτήν την μελέτη όσον αφορά τις αξίες της Ένωσης και κυρίως για το πώς θα εξασφαλίσουμε, πώς θα καταστήσουμε στεγανές αυτές τις αξίες σε σχέση και με το κράτος δικαίου, rule of law. Με αυτή μας την μελέτη καλύπτουμε τέσσερις άξονες και θα σας τα αναπτύξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πρώτα πρώτα να σας πούμε για αυτές τις αξίες και στη συνέχεια να μιλήσουμε για τα βασικά μέσα που έχει διάθεση της Ένωση για να εξασφαλίσει την εφαρμογή αυτών των αξιών στην Ένωση και στη συνέχεια πρόκειται να εμβαθύνουμε για το τι έχει γίνει σε συγκεκριμένε περιπτώσει για Πολωνία και Ουγγαρία. Ε, αυτό θα απασχολήσει τον συνάδελφο Λογοθηκαστήγιο, τον συνάδελφο και τελικά προβαίνουμε σε κάποιες συστάσεις κατακλείδη ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτές τις αξίες να τις καταστήσουμε πιο ασφαλείς, πιο στεγανές σε ένα κράτος δικαίου θεμελιώδεις αρχές και άλλες που διατυπώνται στο άρθρο 2 της Συνδικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 2 είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ε, θεμελιώδες, ε, άρθρο και εξηγεί, το οποίο είναι η ταυτότητα ούτω ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει θεμέλιο τρει άρχε κράτο δικαίου, η rule που ενσωματώνει κάποιες ε, έννοιες που έχει θεσπίσει η Σύμβαση της Βενετίας. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρήθηκε ότι είναι προαπαιτούμενο δημοκρατία στο κράτος δικαίου και αυτές οι αρχές όπως οι αξιαθές δικαιοσύνης, εάν δεν συντρέχει, δεν υπάρχει δημοκρατία. Τα είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 16 σε ένα ψήφισμα πρόσφατα και επίσης ε, οι αξίες της κάθε της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα πάντως. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι μέσα έχει ένωση στη διαθέσή τη, ούτω ώστε να παράσχει την εγγύηση ότι αυτέ οι αξίε πρόκειται να είναι ουσιαστικέ, να μην μείνουν ε, νεκρό γράμμα. Και ότι αυτές οι αρχές θα ισχύσουν στην πραγματικότητα. Ε, έχουμε στα, στη διάθεσή μας τρία μέσα τα οποία τα αναφέρουμε στην εργασία, στη μελέτη πρώτα-πρώτα, η διαδικασία του άρθρου 7 της για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει τη διαδικασία με την οποία οι αξίες για τις οποίες συζητούμε αποκτούν χαρακτήρα συνταγματικό. Γιατί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 ένα κράτος μπορεί να ε, αποστερείται κάποιων δικαιωμάτων εάν μέσω του άρθρου 7 διαπιστώνεται ότι δεν έχει τηρήσει, ότι έχει παραβιάσει ε, κατά συρροήν αυτές τις αξίες. Και έχουμε εδώ πέρα δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση ε, με τρία πέμπτα το Συμβούλιο και με σύμφωνα με το Κοινοβουλίο θα πρέπει να διαπιστώσει ότι υπάρχει κίνδυνος ε, παραβίασης σοβαρής ε, και επίσης μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει πλέον ε, κίνδυνος παραβίασης αλλά υπάρχει καθ' αυτή η παραβίαση των λόγω αξιών και επομένως σήμερα τη διαδικασία του άρθρου 7 Έχουμε ε, ήδη γεγονό την εφαρμογή του. Η Πολωνία και η Ουγγαρία τέλο πάντων άρχισε η εφαρμογή του για να είμαστε πιο ακριβόλογοι. Έγινε με αυτόν με πρωτοβουλία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπή ε, του, 20 17, τότε το άρθρο 7 και ίσχυσε για την Ουγγαρία και στις 12 του, του 18 ενέκρινα το σχετικό ψήφισμα το Κοινοβούλιο και επισημάθηκε ότι υπάρχει κίνδυνο σοβαρή παραβίαση των, άρθρων, των αξιών του άρθρου 2 από την φράση τη Ουγγαρία. Και επίση έχουμε. Ε, έχουμε ήδη πρωτοβουλία για απολός του Συμβουλίου, πρωτοβουλία της Επιτροπής, αυτά στο Συμβούλιο, ακριβώς ε, για κάποιους ε, νόμους που έχουν θεσπίσει αυτές οι χώρες και έχουν σχέση με την δικαιοσύνη και ότι αυτό αποτελούσε πλήγμα στην εξαρτησία της ε, δικαιοσύνης. Ο συνάδελφος θα σας τα πει ενδελεχέστερα στη συνέχεια. Τώρα, δεύτερο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπερασπίσει τις λόγω Η γνωστή διαδικασία επί παραβάση. Τα άρθρα 258 επόμενα τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά τα πράγματα. Διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει παραβίαση τη υποχρέωση που επιτάσσει η συνθήκη σε κάποιο κράτο μέλο. Οπότε προσφεύγει ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από κάποιε προδικαστικέ ε, κινήσει. Οπότε Εάν διαπιστώνεται ότι όντω συντριχεί παραβίαση, καταδικάζεται το κράτο μέλο να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου. Και αυτό ήδη έχει γίνει για την Πολωνία. Πρόκειται για την πιο επιτυχή διαδικασία που έχει ισχύσει για την Πολωνία. Απαιτήθηκε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση του Οκτωβρίου του 18 για την Πολωνία. Και υποχρεώθηκε με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ΔΕΚ το να θέσει εις, ε, ε, εις ε, συνταξιοδότηση 20 συγγνώμη, να, να, να ανακαλέσει από τη σύνταξη 20 τόσους δικαστές των τότε δικαστηρίου. Ε, δικαστές που τους είχε βάλει στη σύνταξη. Βλέπουμε επομένω ότι εφαρμόστηκε το μέτρο, διότι κατόπιν τη αποφάσεω του ΔΕΚ διόρθωσε η Πολωνία και ανεκάλεσε από τη σύνταξη αυτού του δικαστέ. Διόρθωσε αρχική απόφαση. Υπάρχει επίση και το λεγόμενο rule of law framework, δηλαδή η διαδικασία του κράτου δικαίου ε, αυτό το πλαίσιο κράτου δικαίου που θεσπίστηκε το 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μια διαδικασία διαλόγου ούτω ώστε να αποφευχθεί το άρθρο 7 που είναι πολύ πιο αυστηρό και έτσι γίνεται κάποιος διάλογος όταν θεωρείται ότι υπάρχει κάποια συστημική απειλή ε, κατά των θεμελιωδών αξιών και όταν υπάρχουν περιθώρια διορθωτικών κινήσεων. Έγινε αυτό και αυτό για την Πολωνία. Ε, όμως ε, δεν είχε έρθει ο πέρας, οπότε η Κομισιόν κατέφυγε στην διαδικασία του άρθρου 7. Άρα έχουμε αυτά τα μέσα στη διάθεσή μας και τα τρία αυτά μέσα έχουν εφαρμοστεί για την Πολωνία και το άρθρο 7 το οποίο υλοποιήθηκε, το οποίο εφαρμόστηκε για την Ουγγαρία που θα σας τα πει ο συνάδελφος εν τέλει. Τώρα να σας πω τι γίνεται με τις συστάσεις ε, τις οποίες διατυπώνουμε στη μελέτη μας. Εκεί εξηγούμε κατά λεπτός τις προτάσεις, τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των τελευταίων ετών. Ας πούμε, κατά τον 21ο αιώνα ε, έχουμε την πρόταση του Κοινοβουλίου για τη Συμφωνία για Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χειμεροδικαιώματα, ε, καλύφθηκε εκεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε έχουμε λόγω προτάσεις που είναι πολύ αξιόλογες από το Κοινοβουλίο και Κομισιόν. Όμως υπάρχουν δύο ενστάσεις, δύο προβλήματα για αυτές τις προτάσεις. Πρώτα-πρώτα, όταν δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση για τροποποίηση των συνθήκων, τότε αυτά τα θεσμικά όργανα ε, δεν κάνουν, δεν, δεν, μπορούν, δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από ό,τι ισχύει τώρα. Οπότε όταν υπάρχει πρόταση τροποποίησης, ε, φυσικά δεν είναι εύκολο να γίνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις, αλλά τη σήμερα ημέρα ε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολη η τροποποίηση σήμερα. Πάντω υπάρχουν δύο προτάσει που δεν ε, προποθέτουν τροποποίηση των θεμελιωδών συνθήκων. Μία πρόταση λέει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να προσυπογράψει την Σύμβαση των Δικαιωμάτων όπως λέει το άρθρο 6 της ε, Σύνδεξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη πρόταση που είναι πιο σημαντική κατά τη γνώμη μου και αφορά το άμεσο μέλλον ε, σχετικά με οικονομική κύρωση κατά κάποιου κράτους το οποίο έχει παραβιάσει το άρθρο 2. Όμως αυτό θα πρέπει να είναι στοχευμένο. Ε, δεν επιβάλλεται αυτή η οικονομική κύρωση εάν δεν έχει διαπιστωθεί η παράβαση ε, και να έχει διαπιστωθεί η παράβαση είτε μέσω του άρθρου 7 ή μέσω απόφασης του 10. Επομένως, με αυτή την οικονομική κύρωση είναι δυνατόν κάποιο κρατός μέλος να καταδικαστεί. Κατόπιν μη τηρήσεις των υποχρεώσεων που επιτάσσουν οι συνθήκες ή όταν το κράτος αυτό έχει ε, κάνει κάτι που αντιβαίνει θεμελιώδεις αρχές και το κράτος δικαίου. Και έχουμε το άρθρο 322 παράγραφος 1 εδάφιο α για ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή η πρόταση διαφοροποιείται από έναν ε, κανονισμό ο οποίος τώρα σχεδόν ολοκληρώνει τη διαδρομή τους. Αυτόν τον κανονισμό προβάλλεται το ότι μπορούμε να έχουμε ε, χρηματική ποινή που να συνίσταται ε, την αποστέρηση κάποιων, ε, ε, κάποιων πόρων συνοχής που θα πήγαιναν σε αυτό το κράτος. Γιατί προϋποθέτει το ότι οι αποφάσεις ή, ή τέλος πάντων το, το να πλήσει κάποιο κράτος γενικευμένα το κράτος δικαίου, θα πρέπει αυτά λοιπόν αυτές οι πράξεις να στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων ε, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς δεν ενεργοποιούνται αυτές οι κυρώσεις. Αλλά τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που εξηγήσαμε, δεν προϋποτίθεται κάποιο είδους τέτοια βλάβη των οικονομικών συμφερόντων γιατί όταν μιλούμε για παράβαση του άρθρου 2 που οδηγεί στη χρηματική ποινή και έτσι έχουμε τα όσα επιτάσσει το άρθρο 222 παράγραφος 1. Αυτά λέμε στη μελέτη μας, ε, δεν έχουμε πούμε τίποτα άλλο, με ευχαρίστηση σας τα παρουσιάσαμε, αλλά για να ολοκληρώσουμε θα πρέπει να σας πει τις λεπτομέρειες του τι έγινε με την Πολωνία. Να σας τα πει ο Λόπεθ Καστίγιο, συνάδελφος. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Λόπες. Έχετε το λόγο κύριε Καστίλιο. ευχαριστώ. Θα μιλήσω για το ζήτημα τη Ουγγαρία και τη Πολωνία ε, για τα, τις οποίες έχουν ακουστεί πολλά θέματα, πολλά, πολλά, πολλές παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω να εξάγω κάποια συμπεράσματα και κάποια, ε, κάποια αξιολόγηση σε σχέση με τις πρώτες ενέργειες που έχουν αναλυφθεί σε σχέση με την Ουγγαρία και την ε, Πολωνία, γιατί το ζήτημα δεν είναι απλό. Δεν έχει σχέση μόνο με αυτές τις δύο χώρες, αλλά με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι επιπτώσεις είναι, θα είναι, μπορούν να είναι σημαντικές για το μέλλον. Επομένως το ζήτημα δεν είναι η εξέλιξη της συγκεκριμένης διαδικασίας που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά να τη δούμε αυτήν στο πλαίσιο της και τι μας δείχνει για τα, τα όρια που έχει η προστασία των, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις σε ορισμένα κρατή-μέλη. Σε ορισμένα κρατή-μέλη αυτά είναι πιο έντονα, έντονες αυτές οι τάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται στην Πολωνία και στην Ουγγαρία σε αυτές τις ε, περιπτώσεις. Δεν έχουμε μόνο μια υποχώρηση των συνταγματικών ε, χιγγείων, αλλά είναι ευρύτερο το πρόβλημα. Έχουμε να κάνουμε με κόμματα ή τάσεις λαϊκιστικές, ότι έχουμε πλέον κόμματα λαϊκιστικά τα οποία παίρνουν διψήφια ποσοστά, συμμετέχουν στις κυβερνήσεις. Και αυτό δείχνει και πόσο δύσκολο είναι να ακολουθείτε μια διαδικασία με βάση το άρθρο 7 της συνθήκης. Είναι δύσκολο να, να δικαιολογηθεί πολιτικά μια τέτοια πρωτοβουλία. Και επίσης τελικά πρέπει να είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς σε ποιο βαθμό μπορεί να ελέγχει αυτά τα προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα ζητήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη τα οποία τίθεται στο στόχαστρο επικαλούνται την ε, αυτονομία τους ε, στην επίλυση των συνταγματικών θεμάτων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ε, ότι είναι μια κοινότητα δικαίου και αυτό το έχει επαναβεβαιώσει πολλές φορές, έχει αναφερθεί και από το, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασισμένη στο δίκαιο και προσπαθεί να εφαρμόζεται αυτό το, αυτές οι κοινέ αρχές να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την επικράτειά της και αν αυτό δεν συμβαίνει βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν λοιπόν από αυτή την ε, σύντομη εισαγωγή. Θα έρθω πιο συγκεκριμένα στις δύο περιπτώσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε αυτά που ανέφερα στην εισαγωγή και πιο αναλυτικά μετά. Για... Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να δούμε το άρθρο 2 για τις θεμελιώδες αρχές σε, σε, μαζί με το άρθρο 4 της συνθήκης συνδυασμό με το άρθρο 4. Ας δούμε λοιπόν έχοντας υπόψη μας ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχουμε και παλαιότερες αντίστοιχες υποθέσεις το 2000 με την Αυστρία όπου υπήρξε μια προσπάθεια ελέγχου σε πολιτικό επίπεδο Και σε άλλα κράτη υπήρξαν δυσκολίες ή προβλήματα, στην Ιταλία για παράδειγμα. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω με την παρέμβασή μου είναι ότι το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο και δεν αφορά μόνο αυτές τις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, αυτές τις δύο χώρες. Η διαφορά που υπάρχει κατά την άποψή μου μεταξύ της, της περίπτωσης της Πολωνίας και της Ουγγαρίας είναι η εξής για την περίπτωση της Πολωνίας. Το πρώτο που διαπιστώνει κανείς είναι ότι τα πράγματα κινήθηκαν γρήγορα μετά από μια σημαντική πολιτική αλλαγή που συνέβη στη χώρα και είχαμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με πολύ βασικές αρχές του συντάγματος, τη συνταγματικής τάξης. Και ουσιαστικά δηλαδή τη διάκριση των εξουσιών μεταξύ της κυβέρνησης και της εκτελεστικής εξουσίας και της νομοθετικής εξουσίας και της δικαστικής εξουσίας. Και η προσπάθεια ήταν δηλαδή εδώ να διασφαλιστεί αυτή η ουσιαστική διάκριση των εξουσιών και πιο συγκεκριμένα να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ για την Πολωνία βεβαίω μιλούμε για την ε, ανεξαρτησία του συνταγματικού δικαστηρίου. Και σε διάφορα ψηφίσματά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καν, γίνονται αναφορές, μικρές βέβαια, αλλά γίνονται αναφορές στην ανάγκη που υπάρχει για να λειτουργεί το κράτος δικαίου να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των οργάνων του, πολι... του πολιτέματος, του κράτους. Σε ένα ε, για να δημιουργηθεί λοιπόν μια συνταγματική τάξη πρέπει να υπάρχουν όρια στις αρμοδιότητες των εξουσιών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα έχει αναφερθεί και στην ανάγκη καλής συνεργασίας. Αυτό το θεωρώ σημαντικό και εγώ θεωρώ ότι είναι ταυτόχρονα μία απέτηση αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα όριο στο, σε αυτήν γιατί κάθε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επικαλεστεί και την συνταγματική του αυτονομία, δηλαδή το δικαίωμά του να καθορίζει μόνο του τη συνταγματική του τάξη. Δεν μπορεί, θα, θα πει δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μου υπαγορεύει πώς θα καθορίσω τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα μου. Και το ζήτημα αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την Πολωνία, είναι ένα ζήτημα που ανακύπτει και σε άλλες περιπτώσεις άλλων κρατών μελών. Στην περίπτωση τώρα της Ουγγαρίας, οι εξελίξεις ήταν διαφορετικές και πιο περίπλοκες. Ε, έχουμε, τα, τα προβλήματα ξεκίνησαν από το 2011, ως αποτέλεσμα και πάλι μιας πολιτικής αλλαγής, αλλά όχι μόνο. Αλλά εδώ οι εξελίξεις είναι διαφορετικές από την Πολωνία, γιατί έχουμε μια νομοθεσία διαρκής. Ε, ε, πολλές νομοθετικές αλλαγές και επίσης μια συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό ξεφεύγει από το συνηθισμένο πολιτικό διάλογο. Και αγγίζει πλέον ζητήματα που έχουν σχέση με την εθνική ταυτότητα ή επίσης και τη συνταγματική ταυτότητα του κράτους. προσπαθούν στην Ουγγαρία να προσαρμόσουν, λένε, το σύνταγμά τους σε μια συγκεκριμένη εικόνα για την εθνική τους ταυτότητα. Και αυτό έχει σχέση με μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει στη χώρα ε, πολύ πιο πριν. Και υπ' αυτή την έννοια πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της συνταγματικής αλλαγής και αυτών των εξελίξεων που έχουμε διαπιστώσει στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια. οι θεμελιώδες αρχές, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι το οποίο ζητούμε να προσπιστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Και προ... η προάσπιση αυτών γίνεται και μέσω των, συντα... των εθνικών συνταγμάτων. Το οποίο σημαίνει ότι οποτεδήποτε υπονομεύονται οι ε, τα συνταγματικά εχέγγυα που υπάρχουν σε κάθε κράτο μέλο. αυτό υπονομεύει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο σύνολο τη Ένωση. Άρα σημαίνει αυτό ότι υπάρχουν όρια στη συνταγματική αυτονομία των κρατών μελών. Τα όρια αυτά είναι, το όριο αυτό είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και όρια στην εφαρμογή του άρθρου 7 ε, Επίση, υπάρχουν άλλε δυνατότητε. Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει μια προσφυγή ενό κράτου εναντίον ενό άλλου κράτου μέλου στο, στο δικαστήριο. Θεωρητικά αυτό υπάρχει, αλλά είναι πολύ απίθανο. Μας δείχνουν λοιπόν τα όρια το, του μηχανισμού που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές οι δύο περιπτώσεις του, ε, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι θα πρέπει να δούμε το άρθρο 2 της συνθήκης σε συνδυασμό με το άρθρο 4. Ε, γιατί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται και στο εσωτερικό επίπεδο, στο επίπεδο της εσωτερικής συνταγματικής τάξης και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα. Γι' αυτό, όπως έλεγα, όταν υπάρχει μια υπονόμευση της συνταγματική τάξης στο εσωτερικό μιας ε, χώρας, ενό κράτου μέλου, αυτό δημιουργεί υπονόμευση τη της των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο σύνολο τη Ένωση. Γίνεται κατά μία έννοια ένα συνταγματικό πρόβλημα της Ένωσης συνολικά. Και ολοκληρώνω με μια αναφορά στην πρόταση που έχει γίνει. Έχει αναφερθεί σε κάποια από τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να θεσπιστεί τι αυτή η υποχρέωση που πρέπει να έχουν τα όργανα του των κρατών, αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτό έχει αναφερθεί στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σόπφλιν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους ε, δύο καθηγητές που ήρθατε σήμερα. Έχω αρκετές ερωτήσεις και για τους δυο σας. Και θα ξεκινήσω με την πρώτη. Ε, αυτά που είπατε είναι νομική εκτίμηση ή πολιτική εκτίμηση, διότι κατανοώ πως υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην νομιμότητα και την πολιτική. Και αναφέρεστε σε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία είναι πολιτικές πράξεις, οι οποίες έχουν προκύψει ε, από την πολιτική βούληση και όχι απαραίτητα από κάποιο νομικό κείμενο. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω αν έχουν τη βαρύτητα για να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Επίσης, θεωρείται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ενιαίο χώρο νομικά. Και εφόσον ναι, υπάρχει διακρίση ανάμεσα στις παλιές χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, Έπειτα υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή ε, του ενωσιακού δικαίου στα κρατημέλη. Διότι ε, όλα τα προβλήματα στα οποία αναφέρεστε ε, αφορούν χώρες που προσχώρησαν μετά το 2004 τα νέα κρατημέλη. Επίσης παρατηρείται παρεκκλήσει σε ό,τι αφορά τις νομικές πρακτικές. Θα γνωρίζετε φαντάζομαι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των συνταγματικών δικαστηρίων σε αρκετά όπου οι αποφάσεις των συνταγματικών ε, δικαστηρίων ε, αγνοούνται από τα ανώτατα δικαστήρια. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα των νέων χωρών, ε, των νέων κρατών μελών, αλλά προϋπήρχε. Κύριε Καστίγιο, η συνταγματική ταυτότητα στην οποία αναφερθήκατε είναι κάτι το πολύ δύσκολο ως έννοια και σίγουρα γνωρίζετε να μου απαντήσετε ε, την εξής ερώτηση. Ποιος είναι ο μέσος όρος, ποια είναι η διάταξη, η ενάρχηση ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ορίζεται αυτή. Αναφερθήκατε στα συνταγματικά δικαστήρια που έχουν διάφορα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, σε αυτά συνυπολογίζεται και το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, διότι έχει εκδώσει πολύ σημαντικές αποφάσεις για τα άρθρα 4, μάλλον 5. Τέλος, στην παρουσίασή σας αναφέρεστε σε έναν όρο illiberal, ανελεύθερο, στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Τι εννοείται? Ποια είναι η σημασία που δίνεται σε αυτόν τον όρο. Έχει να κάνει με απλή διαφωνία, με την ε, ευρωπαϊκή αντίληψη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή με κάτι άλλο παράνομο. Θα ήθελα τις απαντήσεις σας λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας επισημάνω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επιστημονική συμβολή. Πρόκειται για πρόβλημα πολιτικό, πραγματικό και σοβαρό που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Τα είπε ο Λόπεθ Καστήλιο. Πρόκειται για... Πώς σας το πω κύριε Σόβλη, δεν θα σας δεν σας άρεσε και τόσο πολύ ότι πρόκειται για μια απόπειρα, για, πρόκειται για μια απόπειρα βολής κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο θίγει το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το σύνολο του κράτους του Υγείου που έχουμε οικοδομήσει τελευταία. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το άρθρο 2. Άρα, πρώτα πρώτα. Ευχαριστούμε αυτούς που ανέδεσαν τη μελέτη, αλλά φυσικά ευχαριστούμε και τους δύο καθηγητές που έκαναν, που συνέγραψαν τη μελέτη. Το είπε ο κύριος Σεύλιν Μέρη, ότι υπάρχουμε τώρα μία σύγκρουση, μία αντίφαση εσωτερική στη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ότι πάντοτε θεσπίζονται κάποιοι κανόνες που αφορούν τη διακυβερνητική λειτουργία. Μια που, όπως όλοι γνωρίζουμε, το άρθρο 7 είναι μια πυρηνική βόμβα που βέβαια ποτέ δεν ρίχνεται. Ξέρουμε ότι ακόμα και αν εμείς επικαλεστούμε το άρθρο 7, ποτέ δεν συμφωνήσει το Συμβούλιο λόγω πολιτικών συμφερόντων, λόγω διακυβερνητικών συμφερόντων. Άρα, η επόμενη σκέψη είναι η αναγκαιότητα να βρούμε άλλους μηχανισμούς. Οπότε, να μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε και μέσω του ΔΕΚ για την Πολωνία όσον αφορά την υποχρεωτική συνταξιοδότηση εκείνων των ανωτάτων δικαστών. Άρα έχουμε τώρα δύο θέματα που είναι πολύ σημαντικά. Πρώτα πρώτα την ε, προσήλωση στην ε, Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιώματα όπως το άρθρο 7 κλπ. Άρα έχουμε τώρα τις αποφάσεις του ΔΕΚ σε σχέση με αυτή την ε, ε, σύμβαση. Προσχώρησε και άρα εφαρμογή του 6. Όμως έχει εμπλακεί αυτή η διαδικασία. Τέλη Φεβρουαρίου θα συντηθεί η Κομισιόν με το δικαστήριο. Και κάποιες ενστάσεις του δικαστηρίου δεν μπορούν να παρακαμφθούν. Δεν ξέρω, πρόκειται ποτέ να εφαρμόσουμε το άρθρο 6. Ήδη πάνε 6 χρόνια που προσπαθούμε και δεν καταφέρουμε. Επίσης, αυτό το οποίο ακόμα είναι μέσω της Επιτροπής να έχουμε αυτόν τον ε, κανονισμό, ούτως ώστε να αποστερήσουμε από το κράτος μέλος το επιλήψιμο κάποιους πόρους άμεσο, αποτελεσματικό ε, άρα να το κάνουμε, να το δώσουμε περιεχόμενο. Επίση, κύριε Γκαρίδο, ποια είναι η νομική βάση για την επίκληση του κανονισμού και ούτω ώστε να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση της ε, βλάβης οικονομικών συμφερόντων που φέρνει την ενεργοποίηση των κυρώσεων και του κανονισμού. Μια που ναι, είναι πόρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν να προσθέσουν το κράτο μέλο, αλλά του πόρου του έφεραν τα κράτη-μέλη. Πώ θα γίνει τόσο ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό εργαλείο στα χέρια μα, τι είδαμε στο μεταναστευτικό αυτή την ε, ξεκαθαρή έκφραση των ενστάσεων των κρατών μελών έναντι των συλλογικών αποφάσεων. Και είπαμε ότι μπορούμε να έχουμε θέματα δημοσιονομικά και άλλα. Ε, και γι' αυτό αυτό το οποίο θέλουμε τώρα είναι να δούμε εάν μπορεί η Ένωση να έχει έναν αρκετά αποτελεσματικό μηχανισμό για να καταφέρει. Άρα αυτό είναι το ερώτημα. Τι θα πρέπει να βάλουμε στον κανονισμό που τώρα συζητείτε και διεκπεριώνεται σε Κομισιόν και Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να τον κάνουμε αποτελεσματικό για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Σπινέλη. Grazie, Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους δύο μιλητές. Και όσους έλαβαν το λόγο στη συνέχεια. Να σας πω για τη δική μου εμπειρία. Από όλα τα θέματα που αφορούν Πολωνία και Εγκορία και το κράτος δικαίου. Είχα πάει σε μια αποστολή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στην Πολωνία και η εντύπωση που αποκόμισα, ιδίω στην Πολωνία, είναι η έντονη αίσθηση του ανήκει σε ένα κοινό δικαϊκό χώρο στην Ευρώπη. Όμως, υπάρχουν οι γνωστές ενστάσεις για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 και όλα αυτά, όλη αυτή η προβληματική για το άρθρο 7 θεωρείται ότι είναι αλυσιτελής, είναι φορτισμένη πολιτικά και πέφτει στο κενό τελικά η προσπάθεια εφαρμογής αυτού του άρθρου. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι γίνεται με τις διαδικασίες επί παραβάση και ποιος είναι ο ρόλος του ΔΕΚ. Οπότε, για πέστε μας, κύριοι καθηγητές, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Πώς βλέπετε όλη αυτή την επιφυλακτικότητα έναντι του 7. Και συγκεκριμένα, πώς βλέπετε αυτό, τον, αυτό το σύμφωνο για τη δημοκρατία, ε, το κράτο δικαίου και θέματα δικαιωμάτων που εγκρίναμε εδώ στο Κοινοβούλιο ως εναλλακτική ή συμπλήρωμα του 7. ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφορτήσουμε κάπως πολιτικά το 7 και να αποκτήσουμε πιο το λιγότερο τιμωρητικό εργαλείο. Τώρα όσον αφορά τις ε, οικονομικές κυρώσεις, για πετε μας τι γίνεται. Γιατί εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Ο κόσμος να πληρώσει την ύφη για τα αμαρτήματα των κυβερνήσεων το, το τελευταίο. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον όσα είπατε για το άρθρο 2 σε σχέση με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της συνθήκης. σε σχέση με τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών. <coughs> Γιατί υπάρχει κάποια τέτοια ε, παράδοση. Και επίσης υπάρχουν κάποια άρθρα ευρωπαϊκά ούτως υπήν. Τα λέει και το γερμανικό σύνταγμα στο άρθρο 11 και αφορά αυτή την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και καθορίζει ποιες είναι προποθέσεις για την εκχώρηση αυτή της κυριαρχίας. Για πέστε μου. Τι γίνεται όταν ενεργοποιείται κάποια κοινοτική, ευρωπαϊκή ούτως διάταξη, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με τις εν λόγω διατάξεις των εθνικών συνταγμάτων. Ε, thank you, Enrique Guerrero. Σας ευχαριστώ είχα ζητήσει το λόγο για να μιλήσω για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία είχε παρακολουθήσει η Επιτροπή μας από την αρχή. Είχαμε παρακολουθήσει ο κύριος Σαχαρογή την προηγούμενη θετία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το θέμα. Αλλά με κάλυψαν αυτά που είπε ο Ραμόν, επομένως σας ευχαριστώ, δεν χρειαζόμουν το λόγο. Να έχουμε περισσότερο χρόνο για να ακούσουμε τις απαντήσεις. Uh, Συνάδελφοι, Μερσέδες, αν όχι, θα ήθελα και εγώ να θα κάνω μια ερώτηση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το συμπέρασμα από την έκθεσή σας δεν θα προκαλέσει έκπληξη σε κανέναν μας, ότι δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας τα απαιτούμενα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις συστηματικές απειλές στο στο δικαίου. Μιλήσατε για την χρήση του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 4. Σε γενικέ γραμμέ όμω, ξέρετε, τα προβλήματα αυτά βρίσκονται στο εσωτερικό των κρατών μελών, όχι μεταξύ κρατών μελών. Και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αποτελεσματική στο να αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα των κρατών μελών και δεν ήταν και ο σκοπό τη δημιουργία τη από την αρχή. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, τις οποίους δεν αναφέρατε, γιατί δεν είναι τόσο νομικά ισχυροί, ίσως το 258 ή και άλλοι, το 257. Ε, σε πολλές... Πρώτα απ' όλα έχουμε τα κριτήρια της ένταξης, τα οποία είναι ξεκάθαρα και τα οποία δεν θα πρέπει να τίθενται να αμφιβολώ αργότερα, μετά την ένταξη δηλαδή μιας χώρας. Αν δεν απατώμε υπάρχει και ένας μηχανισμός ε, επαλήθευσης τον είχαμε ονομάσει, τον οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Έχουμε επίσης αιτήσεις εκθέσεις επί τη βάση της ε, εφαρμογής της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχουμε επίσης την αιτήσια έκθεση της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Βιέννη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έχει προτείνει να ενοποιηθούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και όλες αυτές οι εκθέσεις. Αυτή ήταν η δική μας πρόταση, όμως τα άλλα θεσμικά όργανα δεν συμφώνησαν. Αν δεν απατούμε επίση στο Συμβούλιο, μια φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο συζητάει ζητήματα κράτους δικαίου. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας θέσω, πέρα από όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις που τέθησαν και τα επιχειρήματα τα πολύ χρήσιμα που εκθέσατε, είναι το εξή. Στο σύστημα του ΟΗΕ υπάρχει μια τακτική επισκόπηση όχι μόνο του κράτους δικαίου αλλά γενικότερα της ποιότητας της διακυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα αξίζει να έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό να έχουμε ένα μηχανισμό δηλαδή τακτική αξιολόγηση και τη ποιότητα τη διακυβέρνηση και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο μέλλον. Είναι μια σκέψη. Να το προσθέσουμε δηλαδή αυτό πέρα από τα οικονομικά ε, εργαλεία, γιατί κατά την άποψή μου, εντάξει, τα υποστηρίξαμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια μορφή εκβιασμού. Δεν πρέπει να ε, τίθεται έτσι το ζήτημα ε, όταν μιλούμε για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το ζήτημα είναι πολύ πιο σοβαρό, δεν μπορεί να επιλύεται μέσω προστήμων ή της απειλής τους. Δεν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε, μήπως θα έπρεπε λοιπόν στο μέλλον να δημιουργήσουμε ένα σύστημα περιοδικού ελέγχου των κρατών μελών, το οποίο να αξιοποιήσει και τις υφιστάμενες εκθέσεις. Θα δώσω το λόγο στους δύο καθηγητές. Ε, συμφωνήστε μεταξύ σας ποιος θα πάρει το λόγο πρώτος. Ο κύριος Γαρίδο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις μου μου απευθύνθηκαν και μετά θα πάρει το λόγο και ο συνάδελφος για τις υπόλοιπε που είχαν περισσότερο σχέση με τη δικιά του παρέμβαση. Θα απαντήσω με τη σειρά των ομιλητών. Ο πρώτος ε, ομιλητής με ρώτησε αν αυτή η διαδικασία του άρθρου 7 ή και οι άλλες είναι μια αξιολόγηση που γίνεται με νομικούς ή πολιτικούς όρους. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ε, συνδυάζονται αυτά τα δύο, είναι και τα δύο μαζί. Το άρθρο 7, για το άρθρο 7 μάλλον, γίνεται μια πολιτική αξιολόγηση της λειτουργίας του κράτους δικαίου σε ένα κράτος. Για να γίνει όμως αυτή η αξιολόγηση συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλέκονται στο άρθρο 7 και αυτό ε, δίνει πολιτικό χαρακτήρα γιατί έχουν όλα τους, όλα αυτά τα θεσμικά όργανα πολιτικό χαρακτήρα. Όμω τι κάνουν αυτά τα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο του άρθρου 7. Πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσο συστηματικά α, τηρούνται οι αρχές του κράτους δικαίου σε, μια, σε ένα κράτος μέλος. Και λαμβάνουν δηλαδή μια απόφαση πολιτικού χαρακτήρα η οποία μπορεί να έχει συνέπειε, μπορεί να έχει για παράδειγμα τη συνέπεια την αποστέρηση των δικαιωμάτων που κανονικά έχει το κράτο μέλο επί τη βάση των συνθήκων. Αυτό όμω είναι πολιτικό. Το... Όμως το, το γεγονός ότι το άρθρο 7 ε, δίνει τη νομική βάση για να λειτουργεί αυτή η πολιτική διαδικασία, την καθιστά και μια διαδικασία νομική. Επομένως θα έλεγα ότι είναι, ε, ε, ε, ο πολιτικός χαρακτήρας είναι πολύ σημαντικός και προκύπτει από το γεγονός ότι συμμετέχουν όλες, όλα τα θεσμικά όργανα και επίσης έχει και υπάρχει και, και μια εγγύηση ότι θα ληφθεί η σωστή απόφαση και η εγγύηση αυτή είναι το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει την όποια απόφαση ομόφωνα. Ρωτήσατε επίση αν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια, ένας ενιαίος ε, δικαιικός χώρος. Ναι, υπό την έννοια των στο πλαίσιο μάλλον των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές τις οποίες όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διακηρύξει ότι σέβονται. Ένα κράτος το οποίο δεν συμμερίζεται αυτές τις αρχές δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα κράτος το οποίο δεν ε, προασπίζει, για παράδειγμα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το, το, το, κράτος δικαίου και όλες τις υπόλοιπες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι θεμελιώδεις αρχές πρέπει να ε, την χάνουν προστασία και τη χάνουν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη. Στην Ευρώπη έχουμε τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από οπουδήποτε αλλού. Ε, και αυτό έχει, αυτή η προστασία έχει δημιουργηθεί και με δικαστικ, δικαιικούς ε, κανόνες. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κοινό δικηγικό χώρος και τέλος υπάρχει και το δικαστήριο του, ε, της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Λουξεμβούργου, το οποίο έχει δημιουργηθεί ακριβώς για την ενοποίηση των διαφορετικών δικαιωτικών χώρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Με ρωτήσατε επίσης για τις ε, ποιοτικέ διαφορές που βεβαίω υπάρχουν ποιοτικέ διαφορές ανάμεσα στα ε, συνταγματικά δικαστήρια σε τα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό έχουν, αυτές έχουν προκύψει από την διαφορετική ιστορία. Γι' αυτό όμως το άρθρο 7 αναφέρεται και στη σημασία των κοινών συνταγματικών παραδόσεων το λέει συγκεκριμένα, είναι το προϊόν των κοινών συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών. Και, αυτές είναι οι βασικές, και αυτή είναι η βασική αρχή. Αναζητείται λοιπόν μια συνοχή και πολιτική και δικαιική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέση με την παρέμβαση του κ. Χαρογή. είπατε ότι είναι πολύ δύσκολο τελικά να εφαρμοστεί το άρθρο 7 γιατί θα χρειαστεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Ναι, πράγματι, υπάρχουν δυσκολίε στην εφαρμογή του άρθρου 7, αλλά είναι μια δυνατότητα που υπάρχει. Και ακριβώ επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία εφαρμογής του άρθρου 7, προτείνει η Επιτροπή αυτό που ονομάζει διαδικασία για τον έλεγχο του κράτους δικαίου ακριβώς για να Μάλλον, ακριβώ επειδή δεν λειτουργήσε αυτό ο διάλογο για τη λειτουργία του κράτου δικαίου, χρειάστηκε να ξεκινήσει η εφαρμογή του άρθρου 7 στι αυτέ τι περιπτώσει που χρειάστηκε. Εάν η διαδικασία για το διαλόγου. Ε, ε, ή μάλλον οι διαδικασ... άλλες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η διαδικασία επί παραβάση, θα μπορούσε να έχει ακολουθηθεί. Στην περίπτωση της Πολωνίας είχαμε μια διαδικασία επιπαραβάση η οποία οδήγησε σε ακρόαση στο δικαστήριο και η οποία τελικά οδήγησε, ε, ανάγκασε την κυβέρνηση της Πολωνίας να ανακαλέσει την απόφαση της για την πρόσφατη, ε, την πρόορη μάλλον συνταξιοδότηση των δικαστών του συνταγματικού δικαστηρίου, άρα λειτουργήσε. Εδώ η διαδικασία. Με ρωτήσατε επίση ποια ήταν η νομική βάση για τον κανονισμό που συζητείται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα εγκριθεί. Ήταν το 322. με αυτή τη νομική βάση προτείνει η Επιτροπή να μπορούν να επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε ένα κράτος μέλος το οποίο ε, δεν ε, προσβάλλει τις ε, θεμελιώδεις αρχές. Βέβαια, με κάποιες εγγυήσει. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με απόφαση του δικαστηρίου, είτε όταν έχει ξεκινήσει η διαδικασία του άρθρου 7. Όταν έχει καταλήξει μάλλον η διαδικασία του άρθρου 7, τότε μπορούν να εφαρμοστούν κυρώσεις. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό. Τέλος, σε σχέση με την παρέμβαση της κυρίας Πινέλη. Ε, είπατε κάτι πολύ σημαντικό. εάν δημιουργηθεί ένας μηχανισμός με τον οποίο ένα μέρος των πόρων από, το ταμείο, από τα ταμεία συνοχής δεν θα φτάνουν στις χώρες εκείνες που, που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην πραγματικότητα αυτό θα έχει επιπτώσεις για τους πολίτες αυτής της χώρες. Και αυτό πράγματι έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός έτσι ώστε να είναι το κράτος εκείνο που θα πληρώσει. Ε, γιατί είναι δύσκολο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιληφθούν και να δεχτούν να πηγαίνουν πόροι από τους ίδιους, από τους φορολογούμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτη τα οποία παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και για τη δική σας ερώτηση, κυρία Χούμπνερ, είπατε ότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που ήδη λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγχεται το κατά πόσον γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου. Ναι, πράγματι. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί και πολλές διαδικασίες. Τους αναφέρουμε όλους στην έκθεσή μας και πολύ αναλυτικά. Αλλά Αυτές οι διαδικασίες οδηγούν σε συζητήσεις, σε ελέγχους και δεν έχουν οδηγήσει σε κυρώσεις ή σε συγκεκριμένες αποφάσεις ε, που να, που να έχουν αποτέλεσμα. Κατά την άποψή μας είναι σημαντικό να δημιουργηθούν μηχανισμοί οι οποίοι να έχουν, τη δυνατότητα, να, να, να έχουν πολύ πιο ενισχυμένη δυνατότητα εφαρμογή. Όπω για παράδειγμα αυτό ο μηχανισμό που συζητείται αυτή τη στιγμή, όταν, υπάρχουν ε, όταν αντικειμενικά μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει παραβίαση των αρχών τη Ένωση, να υπάρχουν οικονομικέ κυρώσει. Δεν είναι κατά την άποψή μα αυτό ένας εκβιασμός, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν διαπιστώνεται ότι τίθενται ε, σε κίνδυνο η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια χώρα. Σας ευχαριστώ. Σας πολύ. Θα σας παρακαλούσα να είστε σύντομοι. Ναι, ναι, ναι. Να μην διαταράξω τις εργασίες, λέει ο κ. Καθηγητής. Πρώτα πρώτα σας ευχαριστούμε για όλα όσα είπατε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ε, τι να κάνω, λάβει τον γείτονα να κατέληξε έναν καθηγητή για ε, κάτι που τον καίει και που εξειδικεύεται. Ναι, να στα πω τηλεγραφικά. Λέμε για τις της προγραφές του κράτους δικαίου σε απλουρώσεις ελευθερισμού. Τώρα, από τη μία μεριά έχουμε την ε, κυβερνητική λειτουργία και την ε, λειτουργία την, του, του δικαίου. Επομένως, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μην, ε, να μην αγνοεί κανείς το κράτος δικαίου και στην Ομοσπονδική Γερμανία ε, κύριε τι γίνεται με το, με το Σύνταγμα, το Συνταγματικό Δικαστήριο. Το Γερμανικό Συνταγματικό βέβαια και ήταν ο πρώτος ο οποίος υπερασπίστηκε ε, αυτού του είδους την συνταγματική ταυτότητα όπου το ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε και στην ε, Ιταλίδα ε, να με λίγα λόγια. Τι συμβαίνει. Η ερμηνεία του γερμανικού συνταγματικού για αυτή τη ρήτρα αποτελεί μία ε, ευρεία ερμηνεία πέραν των ε, θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Δεν μιλήσαμε για την ε, ενιολογική ε, εξέλιξη αυτών των όρων, αυτών των δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε τώρα. Όμως, ε, κατά τη γνώμη μου, έτσι είχαμε μία στρέβλωση των όσων ισχύουν. Κυρία Χιούμπνερ, επίσης, τι γίνεται με τα κριτήρια ποιοτικής εφαρμογής του νόμου από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί το ένα κράτος να αναμειχθεί στα στεγματικά άλλου κράτους μέλους, ούτε ε, βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των υπαλλήλων της. Τα συντάγματα, τα εθνικά αποτελούν ε, πυλώνες, στηρίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να μην το ξεχνάει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η βάση, το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το Σύνταγμα, Συνταγματική Λειτουργία των Κρατών Μελών. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση της μελέτης αυτής σχετικά με την ε, κατάσταση σχετικά με την πολέμηση της παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πολύ φοβάμαι ότι το πρόβλημα αυτό θα εξαφανιστεί, γι' αυτό καλό είναι να συνεχίσετε κι εσείς τη μελέτη σας έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση του τι ε, συμβαίνει και πώς ε, λειτουργεί το όλο σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα ολοκληρώσω το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης και έχει έρθει η ώρα για τις ψηφοφορίες. Μπορείτε να ελέγξετε αν λειτουργούν οι κάρτες σας. Grazie Presidente, mi scusi. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θέλω, κυρία Πρόεδρε, όμως, να σας πω κάποιες σκέψεις μου που θέλω να τα ξέρουν σαν πριν την ψηφορία. Με απασχολούν τα θέματα τότε την Πέμπτη. Πρόκειται να... Ναι, σας περιμένω. Περιμένω να χαιρετήσετε τους ομιλητές. Θα ψηφίσουμε την Πέμπτη για την αλλαγή κάποιων ε, διαδικασιών είναι πολύ σημαντικέ, δεν είναι τυπικέ. Θα έχουν επιπτώσει όσον αφορά τη δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου αυτέ οι αλλαγέ που θα ψηφίσουμε. Και σα τονίζω το εξή. 86, 87 και 88 είναι σχετικές τροπολογίες που προέρχονται από τους ε, σοσιαλιστές, λαϊκό κόμμα, ε, φιλελεύθερους συντονιστές. Δεν έχουν ποτέ συζητηθεί στην Επιτροπή μας κόντρα σε αυτά τα οποία προβλέπει το του κανονισμού με αυτές τις τροπολογίες με απλή πλειοψηφία και απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων θα είναι δυνατόν να διαλυθεί, να παρεμποδιστεί η λειτουργία κάποιας πολιτικής ομάδας. Δεν υπάρχει ούτε ένα αντικειμενικό κριτήριο που θα οδηγήσει στην προϋπόθεση, την προαπαιτούμενη δηλαδή του να μην υπάρχει η έλλειψη συνοχής πολιτικής ομάδας για να ενεργοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Όμως έχουμε δύο πολιτικές μεγάλες ομάδες ε, που αποτελούν πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφής η πλειοψηφία που κάνουν αυτές οι δύο πολιτικές ομάδες. Όμως Μα τι γίνεται, από πότε απονευρώνεται η, η αντιπολίτευση σε αυτό το κοινοβούλιο. Έτσι, δεν θα υπάρχει συζήτηση στην Ολομέλεια. Θα πρέπει να ζητηθούν αυτές οι τροπολογίες. Έτσι, έχουμε την τυραννία, τη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ας μου πούν, ας μου το εξηγήσουν αυτό που θέλουν τέτοιες τροπολογίες με έναν τρόπο τόσο οίκιστα διάφανο. Θα πρέπει να αποσυρθούν αυτές οι τροπολογίες. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο. Οπότε παρακαλώ συνάδελφοι όλοι, όλοι δώστε τη μάχη της ε, δημοκρατίας. Όλα αυτά παραβλάπτουν ε, την εκστρατεία μας για τις ε, εκλογές. Πάντως, εμείς θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί έτσι θίγεται ο πλουραλισμός και δημοκρατία στο Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, όσο καταλαβαίνω ήταν μια πολιτική δήλωση την οποία φυσικά και έχει δικαίωμα να κάνετε και χαίρομαι που χρησιμοποιείτε την ευκαιρία ε, που έχετε. Όμως αυτό είναι πέραν των δυνατοτήτων της Επιτροπής ε, η διάσκεψη των Προέδρων θα αποφασίσει για το παραδεκτό των τροπολογιών αυτών. Αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε ως Επιτροπή ΑΦΚΟ να εξετάσουμε το ενδεχόμενο περαιτέρω τροποποιήσεων στην, στον εσωτερικό κανονισμό. Έτσι ώστε να δούμε αν ε, θέλουμε πριν λήξει η θητεία μας να προχωρήσουμε σε αλλαγές ή αν θα τα αφήσουμε για την επόμενη θητεία. Βέβαια, να μην ανοίξουμε τη συζήτηση καλύτερα, αλλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αργότερα. Ναι, ναι, έχετε το λόγο. Ωραία, δεν θα συζητήσουμε, αλλά η παρέμβαση του κύριου το χρήζει απάντηση, διότι μας παρακολουθούν ζωντανά στο διαδίκτυο και ακούγονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ότι δηλαδή θέλουμε να περιορίσουμε τον πλουραλισμό, αυτό δεν ισχύει, δεν είναι αλήθεια. Είμαστε το πιο ανοιχτό κοινοβούλιο στον κόσμο. Οποιαδήποτε πολιτική ομάδα μπορεί να ενωθεί με κάποια άλλη. Αυτό που δεν ε, πρέπει να επιτρέψουμε βέβαια να ξανασυμβεί, είναι μια ψεύτικη πολιτική ομάδα και αυτά τα ε, ψέματα ότι δεν έχουν καμία σχέση, δεν συναντιούνται, δεν έχουν ούτε κοινή πλατφόρμα, ούτε τίποτα. Στην ουσία ε, συστάθηκε μια πολιτική ομάδα για να ε, αποκομίσει τα προνόμια που έχει μια τέτοια από το Κοινοβούλιο. Νομίζω πως αυτή η τροπολογία λοιπόν έχει αξία, πρέπει να είναι εκεί. Κανείς δεν ήταν έτοιμος για τη σύσταση μιας ψεύτικης πολιτικής ομάδας και δεν υπάρχει νομική βάση στον ιστορικό κανονισμό για το πώς ε, μπορούμε να κινηθούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο μετά τις ευρωεκλογέ θα πρέπει να είναι έτοιμο. Να ξέρει τι πρέπει να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Και να ε, ψηφιστεί στην Ολομέλεια με ε, απόλυτη πλειοψηφία για το αν μπορούμε να... Γιατί αν έχουμε μία ουσιαστική πολιτική ομάδα με πολιτικό προσανατολισμό ή μία ψεύτικη ομάδα η οποία έχει συσταθεί με σκοπό το την αποκόμιση κέρδους. Ωραία, μισό λεπτό διακόπτη πρόεδρος. Ε, Μία διευκρίνηση σχετικά με τις ε, διαφορετικές ερμηνείες τη τροπολογία αυτής που κατατέθηκε. Ε, αυτά είπαμε τέλος η συζήτηση. Σας υποσχέθηκα ότι αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε αργότερα. Να περάσουμε όμως τώρα στην ψηφοφορία διότι έχουμε και πρόγραμμα. Πρώτη ψηφοφορία. Δοκιμαστική. Βάλτε παρακαλώ τις κάρτες ε, στο μηχάνημα για να ελέγξουμε αν λειτουργούν. Επίσης, ε, πρέπει να ψηφίσουν και αλλού οι συνάδελφοι, οπότε βιαστείτε. 21 τα μέλη, για να δούμε πώς είναι εδώ. περισσότερες κάρτες λειτουργούν, ωραία. Χρειάζομαι λοιπόν την σύμφωνη γνώμη σας για να εγκριθεί το, η διόρθωση σχετικά με την έκθεση Σπινέλη. Δεν χρειάζεται ψηφοφορία, απλά την συγκατάθεσή σας. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία, λοιπόν, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στη διόρθωση. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ευρωεκλογών. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Τελική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, μία αποχή. Τελειώσαμε λοιπόν. Περνάμε στην έκθεση Σόπφλιν για την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινή δήλωση ε, που διασφαλίζουν κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών. Συμβαστική 1. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην 14. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπατζ 3 υπέρ κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά, badge 4, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. NV8, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Έκον 1 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Ένβη 6 πρώτο τμήμα μόνο υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την NV6. Πέρας. Απορρίπτεται. NV9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 30. Υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές. Είστε υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα, όχι, δεν το ψηφίσουμε. Συμβαστική 10. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Νέα υποπικεφαλίδα, προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ξέρετε, τι ψηφίσετε υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Μπατζ 2. Ε, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Κοντ 10. Υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Μπατζ 6 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Μπατζ 8 και κον 5 είναι ταυτόσιμε. υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Μπατζ 9 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Μπατζ 10 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Κον 2 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. κον 3 υπέρ. Θα ελέγξουμε την ε, κοντ 3. Τε, πέρας, πέρας. Εγκρίνεται. Κοντ 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικό αναφορέ. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστέ είστε υπέρ. Εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά θα ελέγξουμε την τροπολογία 8. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Μάλιστα, 21 ψήφοι ψήφη υπέρ. Όλοι ψηφίσατε υπέρ. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Δεν συμβαίνει συχνά. Α, τι θέλετε να καταψηφίσετε. Όχι, να ευχαριστήσω την Επιτροπή <coughs> όμως που μου ε, υπερψήφισε ομόφωνα την έκθεση. Να ευχαριστήσω λοιπόν και όσους συνεργάστηκαν για την κατάρτιση της έκθεσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω η Επιτροπή έπραξε κατά το δοκούν. Περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία. Ψήφισμα για την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης από τον Ραμόν Χαουρέγγι Ατόντο και από άλλες ομάδες ψηφίζουμε με ονοματιστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεν υπάρχει ομοφωνία σχεδόν όμως 19 ψήφοι υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Νομίζω πως ε, τελειώσαμε λοιπόν εδώ με τις ψηφοφορίες και με τις συνεδρίες της Επιτροπής. Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε στα διάφορα, εκτός αν θέλετε να συζητηθεί κάτι. Ο κύριος Βίλαντ, στο σημείο 10, θέλετε να πείτε κάτι για τα διάφορα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να επιστρέψω στην έκθεση Σόπφλιν, αλλά όχι στο περιεχόμενο, ως προς τον κατάλογο της ψηφοφορίας και να πω ευθέως ότι η προετοιμασία για την ψηφοφορία αυτή με τα χρώματα είναι υποδειγματική. Έτσι όπως φαίνεται τα χρώματα στην σελίδα. Η γραμματεία λοιπόν έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά ε, και ξέρετε, πολλοί από εμά ψηφίζουμε σε διάφορες επιτροπές και είναι πολύ δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ε, προτείνω η κατάλογη ψηφοφορίας να ε, μοιάζουν με αυτόν που λάβαμε για σήμερα, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσει για όποιους ε, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν σε άλλη ψηφοφορία, σε άλλη επιτροπή. Λοιπόν, να ακολουθήσουμε το τη χρωματική διάταξη αυτών των καταλόγων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βίλαντ. Οι συνάδελφοι στη γραμματεία δεν είναι τέλειοι, αλλά πλησιάζουν την τελειότητα. Θα λάβω λοιπόν υπόψη την πρότασή σας. Λύεται η συνεδρίαση. επόμενη συνεδρίαση 20 Φεβρουαρίου, εκτός αν συμβεί κάτι, ελπίζω για καλό, και χρειαστεί έκτακτη συνεδρίαση σας. Ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.